Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις πέρασε το ακαδημαϊκό μας τέταρτο ε, και τηρούμε το ακαδημαϊκό τέταρτο και γενικώ τους ακαδημαϊκούς κανόνες γιατί στην δημόσια κρόασή μας έχουμε και κορυφαίους ε, πανεπιστημιακούς και έγκυρους εμπειρογνώμονες. Όπως ξέρετε, θέμα της σημερινής δημόσιας ακρόασης είναι η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης στην Ευρώπη. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους καλεσμένους εμπειρογνωμονές μας και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Να πω δύο λόγια εν είδη Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι ποικιλόμορφη Ε, και καλό θα είναι να την αξιοποιήσουμε αλλά και να την αναβαθμίσουμε διευρύνοντας το μερίδιο της παραγωγής πρωτεΐνης, φυτικής μάλιστα πρωτεΐνης. Κάτι που εμπίπτει στις δυνατότητες Ευρωπαϊκής Γεωργίας, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής ε, επαρκώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Επανειλημμένω μα έχει απασχολήσει. Και δυστυχώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, παρόλο που μιλούσαμε για την ανάγκη ε, παραγωγή φυτική πρωτενη σε χώρια, ε, δώσαμε στον πειρασμό να εισάγουμε φθηνότερη σόγια από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των φυτικών μας καλλιεργειών, των πρωτεϊνούχων φυτικών καλλιεργειών και γι' αυτό διοργανώνουμε και σήμερα την αυτή δημόσια ακρόαση για να ακούσουμε τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Μάλιστα αυξάνεται και η πίεση από την κοινωνία, από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για μεγαλύτερη παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. το καθένα ξεχωριστά λίγο πριν του δώσω το λόγο. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο καθηγητής Bernhard Σέφερ. Θα μας κάνει την παρουσίαση για τα ψυχαθή καρπό, τις ευκαιρίες της προμήθειας σε φυτική πρωτεΐνη και καινοτόμα καλλιεργητικά συστήματα. Ο κύριος Σέφερ, ο καθηγητής Σέφερ, είναι κορυφαίος εμπειρογνώμονας για το θέμα αυτό από το Πανεπιστήμιο της Νοτιού Βεσφαλίας και είναι και πρόεδρος ε, ε, του Τμήματος ε, Πρωτεϊνικές Καλλιέργειες της Επιτροπής για την Παραγωγή και τη Διαχείριση σε Ελαιούχες και Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες της Ένωσης για την Πρόθεση Ελαιούχων και Πρωτεϊνούχων Φυτών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, για την κτηνοτροφία στην Γερμανική Γεωργική Κοινότητα. Έχουμε κατόπιν τον κύριο Τζέι Γκονσόφσκι, που είναι ε, δόκτωρ ε, γεωργίας και εργάστηκε και σε πολλές διπλωματικές θέσεις, ήταν και πρέσβης και μάλιστα μέρο μόνιμη μόνιμης τη Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σα στο Πανεπιστήμιο Κάρδιναλ Στέφαν Βεσσίας και στην Πολωνία. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι εμπειρογνώμονες του πρώτου πάνελ. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον καθηγητή Σέφερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Σέφερ. Ja, Herr Vorsitzender, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να σας κάνω αυτή την παρουσίαση με το θέμα που μας υπενθύμησε ο Πρόεδρος. Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της ε, παρουσίασής μου. Απαρτίζεται από έξι σημεία. Θα σας μιλήσω πρώτα τις εκτάσεις παραγωγής που είναι χαρακτηριστικές για τις τέσσερις κατηγορίες ε, άρακα, φασόλια, λούπινα, σόγια με επιλεγμένα κράτη-μέλη, όπου είχαμε τα τελευταία χρόνια μειωτική τάση στις καλλιέργειες και μόνο το τελευταίο χρόνο, με τάση που και φέτος, 2015-2016 δηλαδή, ε, σημειώνεται σημαντική αύξηση των ε, καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις μεγάλες αυτές καλλιέργειες. Εν γέννη, οι φυτικές πρωτεϊνικές καλλιέργειες στην Ευρώπη είναι ελληματικές πάντα. Μεγάλο κοινό λοιπόν, περί το 70% σημειώνεται και καλύπτεται από εισαγωγές, κυρίως για τις όγες βέβαια. Άρα έχουμε και μειωμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμες και μεγάλο έλλειμμα με το οποίο ξεκινάμε. Και βλέπετε εδώ ότι αυτές οι καλλιεργήσεις μας εκτάσεις από το 2014 με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ σημειώνει χάρη στο greening το πρασίνισμα μια μικρή άνοδο. Από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν αυτή την παραγωγή καθώς έχουν μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων ε, καλλιεργειών στις ε, εκτάσεις τους. Χάρη και στην οικολογική καλλιέργεια λοιπόν. Και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη άνοδο πρέπει να υποστηρίξουμε τις εκμεταλλεύσεις. Κίνητρο Φερρυπίν. Κίνητρο θα μπορούσε να είναι η ε, ενίσχυση της στάθμισης του παράγοντα πρασινίσματος. Ξέρω ότι είναι ένα 0,7% ε, ε, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα προς ένα η συμμετοχή του ε, τομέα των προτεραινούχων καλλιεργειών στο πρασίνισμα, η στάθμιση του δηλαδή. Επίσης, εδώ έχουμε να κάνουμε με καλλιέργειες που έχουν στόχο την ανθρώπινη διατροφή. Τα πλεονεκτήματα για την υγεία είναι γνωστά και η αίσθηση του κορεσμού και η χαμηλότερη ε, πίεση του αίματος, ε, υποκατάσταση των υδατανθράκων από ε, άλευρα σιτηρών, μείωση της σύνθεσης της χολεστερόλης και κινδύνου καρκινογένεσης και επίσης εξασφάλιση σημαντικών ίχνων στοιχείων και βιταμινών. Και η τάση είναι όλο και μεγαλύτερη γιατί βλέπουμε ότι ζητάει ο κόσμος όλο και περισσότερο φυτική πρωτεΐνη. Ταυτόχρονα. συνέπειες ε, επιπτώσεις εφόσον ε, μπορέσουμε να μειώσουμε και τις εκπομπές των ε, αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή αντικαταστήσουμε την παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης με τον ε, δείκτη εδώ ότι έχει πολύ χαμηλότερη συμμετοχή σε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα ή αερίων θερμοκηπίου και είναι ενεργειακά πιο οικονομική. Άρα έχουμε ένα διτά θετικό αποτέλεσμα και αηφορία της ανθρώπινης διατροφής. Το οικονομικό σύστημα και το σύστημα διαχείρισης των γεών ωστόσο θα μπορούσε και να ωφεληθεί. Εδώ έχουμε μια πειραματική καλλιέργεια με φάβα και και βρώμη. Βλέπετε τις ε, ε, σημαντικές εξοικονομήσεις ακόμη και σε λιπάσματα. Άλλα λοιπόν ωφέλη που βλέπουμε είναι η μείωση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γενικότερα της επεξεργασίας των εδαφών. 25 χρόνια τώρα κάνουμε ερευνησμένα συστήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ θετικές συνέπειες, ε, αηφορία και ενίσχυση της παραγωγικότητας ε, ε, του εδάφους, ε, σημαντική, σημαντικό στοιχείο των, της δομής του εδάφους, ενίσχυση της βιοπικιλότητας, σταθεροποίηση των διαστρωματώσεων του εδάφους και μπορούμε να έχουμε συστήματα Ε, προστασίας του εδάφους χάρη σε ε, παραπροϊόντα των ε, πρωτεϊνούχων, έτσι όπως βλέπετε στη φωτογραφία εδώ, με τη δυνατότητα να αποφύγουμε τα παραδοσιακά λιπάσματα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Και αυτά λοιπόν συμβάλλουν και στην αηφορία και σε ένα σύγχρονο σύστημα γεωργικής παραγωγής. Εδώ μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικές ε, ε, εξελίξεις ως προς την χρήση των θερινών καλλιεργινών αλλά και των χειμερινών. Τώρα τα ωφέλη που καταγράφουμε ιδιαίτερα για την ε, Γερμανία είναι αυτά τα σχετικά με την ε, αποφυγή χρήσεως ε, ζυζανιοκτώνων. Ιδιαίτερα όλων αυτών των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη μεγαλύτερη, στις μεγαλύτερες ποσότητες και οι οποίες πρέπει να περάσουν μέσα από ένα σύστημα επανακαταχώρησης και αδειοδότησης που όμως μπορούμε να ε, απορρίψουμε προκειμένου να αντικαταστήσουμε από ε, ψυχανθή. Έχουμε μπορέσει να αντικαταστήσουμε Ε, ε, πειραματικά ε, ζυζανιοκτώνα, αλλά, μάλλον εντομοκτώνα, αλλά δεν είναι πάντοτε η αγορά πρόσφορη. Ανταγωνιστικότητα λοιπόν χαμηλή, οι τιμές της αγοράς είναι χαμηλές και μερικές φορές δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση σε ορισμένα τμήματα αγοράς ώστε να προσφέρεται το κίνητρο της παραγωγής αβεβαιότητα υπάρχει σε σχέση με τη χρήση των ε, ψυχανθών. Ε, η σόγια είναι μια σταθερή παραγωγή με γνωστή ποιότητα και διαθεσιμότητα. Αλλά υπάρχουν ε, στοιχεία στην αλυσίδα προμήθειας που δεν είναι γνωστά ή δεν είναι αρκετά διαφανή. Αυτό που συνιστούμε θα ήταν απλούστευση και εναρμόνιση της διαδικασίας καταχώρησης των ζανιοκτών που δεν γίνεται de facto για την καταχώρηση των συνεκτώνων. Θα πρότεινα επίσης την ενίσχυση του παράγοντα στάθμισης στο πρασίνισμα, στο greening, στο 1 προς 1. Επίσης προαγωγή νέων αλυσίδων αξίας, ιδιαίτερα για τις καινοτόμες τροφές και θα, προτιμούσα, θα πρότεινα να ενισχυθεί η αντικατάσταση της αγόμενης σόγιας από ε, πρωτεϊνούχες καλλιεργίες ισοδύναμες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον ε, κύριο Γκονσόφσκι, τον καθηγητή Γκονσόφσκι. Θα τον καλούσα στο βήμα. Ε, Σα ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και συγχαρητήρια γιατί ε, επισημαίνετε το τόσο σημαντικό θέμα τη σόγιας και των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών. Υπάρχουν και άλλα θέματα που ε, είναι συναφή με τις εισαγωγέ της σόγιας, όπως το θέμα της ενεργειακής εξάρτησης. Στην περίπτωση των τροφίμων έχουμε κάπως διαφορετικά προβλήματα. Αυτά αφορούν την μεγάλη δημογραφική αύξηση, την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Φαίνεται από την έκθεση της Επιτροπής ότι στις επόμενες δεκαετίες αναμένεται αύξηση της παραγωγής τροφίμων και της προσφοράς μεταξύ 60 και 110%. Θα περάσω τώρα στα τέσσερα σημεία της παρουσίασής μου. Θα ξεκινήσω με τη σημασία που έχουν οι γεωργικές πολιτικές. Και θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση των γεωργικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζίλιας. Εγώ χρησιμοποίησα συνθετικούς δείκτες, δηλαδή είδαμε την, μικτή, ε, την αξία της μικτής γεωργικής παραγωγής. Βλέπουμε εδώ την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βραζιλία από το 1970 μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε ότι στις δύο πρώτες δεκαετίες είχαμε μία αύξηση της ε, μεικτής ε, γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά μία σταθεροποίηση σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Στην περίπτωση της Βραζιλίας διαπιστώνουμε μία σταδιακή και σταθερή αύξηση της ε, μεικτής ε, αξίας της γεωργικής παραγωγής. Τώρα, μια και μιλούμε για τη σόγια, θα δούμε την κατάσταση της σόγιας και όχι μόνο της σόγιας, αλλά και την κατάσταση της βραζιλιάνικης γεωργίας εν γέννη. Η Βραζιλία ήταν γνωστή για πολλές δεκαετίες ως ε, κύριος εξαγωγέας ε, ε, καφέ και ζάχαρης. Στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε ο πρώτος εξαγωγέας βόλου κρέατος, κρέατος πουλερικών και σόγιας. Εμείς όμως ε, ασχολούμαστε κυρίως με τη σόγια. Θα δούμε λοιπόν την παγκόσμια αγορά σόγιας. Φαίνεται από την ε, διαφάνεια αυτή και από το γράφημα του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας ότι η Βραζιλία δεν είναι μόνο υπαριθμόν εξαγωγές ε, σόγια σήμερα, αλλά θα είναι και ο υπαριθμόν Παγκόσμιο εξαγωγές και στο μέλλον. Ας δούμε τώρα τις εισαγωγέ. Όπως βλέπετε, ο κύριος εισαγωγέας ε, σόγιας είναι η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεύτερος εισαγωγέ, με τεράστιες εισαγωγές, όπως ε, είπατε και εσείς στην αρχή, κύριε Πρόεδρε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα με την προσφορά φυτικής πρωτεΐνης. Από τεχνολογίας δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της καλλιέργειας σίτου και της καλλιέργειας σόγιας, γιατί χρησιμοποιούνται τα ίδια μηχανήματα, σχεδόν ίδιες τεχνολογίες. Αν κοιτάξουμε όμως την κατάσταση εκ του σύνεγγης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εξαγωγές σιτήρων, ε, σίτου κυρίως. Και μάλιστα ταυτόχρονα είναι ο δεύτερος παγκόσμιος εισαγωγές σόγιας. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί οι Ευρωπαίοι γεωργοί δεν ακολουθούν το παράδειγμα των Αμερικανών γεωργών που στηρίχθηκαν στις προβλέψεις των τιμών ε, ΣΥΤΟΥ και ΣΥΚΑΛΙΣ ε, στο χρηματιστήριο ε, πρώτων αγαθών του Σικάγο και να μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους από καλλιέργειες ΣΥΤΟΥ σε καλλιέργειες σόγιας. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών διαπιστώνουμε ότι τα επίπεδα απόδοσης ΣΥΤΟΥ και σόγιας στις Ηνωμένε Πολιτείε και στη Γαλλία είναι περίπου ίδιες μεταξύ δεκαετίας του και του 2011. Βέβαια, στο μεταξύ τριπλασιάστηκαν οι αποδόσεις του σε σχέση με τη σόγια στη Γαλλία. Τώρα, αν δούμε τις υπόλοιπες 27 χώρες και συγκρίνοντας ε, τις ε, αποδόσεις της παραγωγής σύτου και των βασικών ψυχανθών, βλέπουμε ότι είναι διπλάσιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες μήπως είναι ορφανές καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την απάντηση τη βρείτε εύκολα στο, στην περσινή εικόνα της Γεωργίας και την αντίστοιχη έκθεση. Έχει μειωθεί η τις τελευταίες δεκαετίες δραστικά η, μείωση, η παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών, κυρίως επειδή δεν είναι ελκυστικά οικονομικά, αλλά και εξαιτία των αδοσμολόγητων ε, εισαγωγών ε, πρωτεϊνούχων και ελαιούχων σπόρων, που ρίχνουν φοβερά τις τιμές. Καταρχήν, η παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών, πρωτεϊνούχων καλλιεργιών. Βλέπετε ότι ε, είναι μειον η εικόνα για τα ψυχαθή και μάλιστα το 1960, πριν την κοινή γεωρική πολιτική, από τότε, από το 1960, ε, μειώνεται η επιφάνεια των αγροτεμαχίων. Μετά την εισαγωγή της κοινή γεωρικής πολιτικής, η επιφάνεια των πρωτενούχων σπόρων ε, μειώθηκε, σε αντίθεση με τη Βραζιλία που αυξήθηκε η επιφάνεια καλλιέργειας πρωτεϊνούχων ε, φυτών, σόγιας και άλλων. Τώρα, γιατί είναι οικονομικό δεν είναι οικονομικά ελκυστικέ αυτέ οι πρωτενούχε καλλιέργειε. Ο Θέοδρο Βίλιαμ Σούλτ, βραβείο Νόμπελ Οικονομικό του 1979, είπε ότι οι γεωργοί μπορούν να μετατρέψουν το χώμα σε χρυσό εφόσον είναι πρόσφορε οι οικονομικέ συνθήκε. Για να δούμε όμω ποιε είναι αυτέ οι οικονομικέ συνθήκε. Το πιο σημαντικό θέμα που επηρεάζει ε, την σημασία τη της σόγιας είναι οι αδοσμολόγητες εισαγωγέ της σόγιας. 65% με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, των ε, των εισαγωγών του 2014 αφορούν τέτοιου είδους ε, προϊόντα, σόγια, πίτες, ελαιούχων σπόλων και ούτω καθεξής. Τώρα για να δούμε την επιρροή της κοινή γεωρικής πολιτικής. Όπως είπε και ο καθηγητής Σέφερ, το τελευταίο καιρό έχουμε κάποιες θετικές αλλαγές, αλλά μικρής εμβέλειας. Βλέπουμε τώρα τα ερευνητικά προγράμματα και τα προγράμματα επέκτασης. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη μα έδωσε τα σχετικά στοιχεία και βλέπουμε ότι ε, τα σχέδια για του πρωτεϊνούχου ε, πόρου ε, είναι λιγότερα από 20 εκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια αντίθετα είναι τα κονδύλια που αφιερώνουν στην έρευνα οι υπόλοιποι εταίροι μας για τις πρωτεϊνούχε καλλιέργειε. Βλέπετε λοιπόν ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργία δεν δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα με τόσο πενιχρά προγράμματα στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων ε, φυτών. Τώρα, ποιε είναι οι προτάσει. Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών με βιολογική διαφοροποίηση, καινοτόμα οικονομικά κίνητρα, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα τη διαφοροποίηση των εισαγωγών μα. Τώρα, βιολογική διαφοροποίηση, το πρώτο σημείο θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα ε, φυτά να καλλιεργούμε. Έχουμε βέβαια διαφορά στο πρωτεϊνικό τους περιεχόμενο, από 14 μέχρι 37%. Αυτές είναι οι διαφορές από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο περιεχόμενο πρωτεΐνης. Ελάχιστη ως μέγιστη περιεκτικότητα πρωτεΐνης. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό και για τους γεωργούς και για τους κτηνοτρόφους να βελτιώσουν την κατάσταση διαφοροποιώντας ε, τις καλλιέργειες και χρησιμοποιώντας πρωτεϊνούχα φυτά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα πρωτεΐνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα συστήματα αποζημίωσης για τη δέσμευση του αζότου. Σε περίπτωση ψυχανθών και οσπρίων, η δέσμευση αζότου αντισταθμίζει τη χρήση λιπασμάτων. Και όπως αναφέρθηκε στην έκθεση της κυρίας Ανθέα Μακκίνταιρ, τα ζωτούχα λοιπάσματα είναι σημαντικά για, την, για τις υψηλές αποδόσεις. Βέβαια, για την Παρασκευή τους χρειάζεται 50% ενέργεια από ρηκτά καύσιμα. Αυτό είναι το 50% της ενέργειας από ρηκτά καύσιμα που χρησιμοποιεί η γεωργία. Οπότε γιατί να παράγουμε τέτοια λοιπάσματα ζωτούχα και ταυτόχρονα να ρηπαίνουμε το περιβάλλον. Αντίθετα θα πρέπει να ενισχύσουμε τις παραγωγές ε, ψυχαθών και οσπρίων. Μέχρι σε ό,τι αφορά την ε, επιβολή δασμών. Αν δεν επιβάλλουμε δασμούς ε, στις αγωγές σόγιας και πίτας από ελέγχους σπόρους, δεν πρόκειται να βελτιώσουμε τη δική μας παραγωγή και το θέμα των καινοτόμων κινήτρων. Αν εξετάζουμε το θέμα από τη σκοπιά των εισαγωγών, γιατί να μην κοιτάξουμε προς τα Ανατολά, προς την Ουκρανία, προς τη Ρωσία, που είναι πιο κοντά μας. Αυτοί οι στενότεροι δεσμοί θα ευνοήσουν όχι μόνο τους γεωργούς μας, αλλά και την οικονομία μας τα συμπεράσματά μου τώρα. Από τεχνολογική άποψη, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ καλλιέργειας ήτου και καλλιέργειας σόγιας. Δεύτερον, η βασική λόγη για το απαράδεκτα υψηλό επίπεδο εισαγωγών σόγιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίστηκαν ως ε, οι ατασμολόγητες εισαγωγές ε, φυτικής πρωτεΐνης, οι χαμηλές αποδόσεις των ε, πρωτεϊνοχών καλλιεργιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλλειψη ε, έρευνας, ε, ενεπαρκής διαφοροποίηση και έλλειψη σαφών πολιτικών αποφάσεων. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί και μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αν και εγώ είμαι κάπως απεσιόδοξος, γιατί δεν υπάρχει δεδηλωμένη και ισχυρή πολιτική βούληση για να επιληθεί το πρόβλημα της έλλειψης ε, φυτικής πρωτεΐνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε κάποιους ακτιβιστές ε, κατά των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Είναι πολύ ισχυρά αυτά ε, τα λόμπι, όπως ισχυρά είναι και τα λόμπι των εισαγωγών, ε, εισαγωγέων σόγιας. Και έχουμε και τους ε, διάφορους, τα διάφορα επίπεδα της κοινής γεωρικής πολιτικής. Και επίσης αδυναμία του, των λόμπι των Ευρωπαίων γεωργών. Είναι ένας από τους άλλους λόγους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα και μάλιστα τήρησε και το χρόνο σας. Όπως είπαμε, αυτό είναι το πρώτο τμήμα της δημόσιας ακρόασης. Μετά τις δύο παρουσιάσεις θα ακολουθήσει η συζήτηση. Πρώτος ζήτησε το λόγο ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ του ομιλητέ μα για τι τόσο ενδιαφέρουσε παρουσιάσει του. Πριν από λίγα χρόνια, σε αυτό το κοινοβουλευτικό σώμα, είχα την ευκαιρία να ακούσω ένα Γάλλο καθηγητή που ονομάζεται Μάρκ Ντιφινιέ, ο οποίο παρότρινε να σταματήσουν ε, οι συμφωνίες Blair House, διότι τότε συζητούσαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο, δηλαδή το 70% των ζωοτροφών μας ερχόταν από τις Πολιτείες, από την Αμερική μάλλον, ΗΠΑ και Βραζιλία. Ε, κατάλαβα από την παρουσίασή σας ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τι συμφωνίε όχι μόνο με τι γειτονέ χώρε, αλλά να κοιτάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει και μια στρατηγική σε σχέση με τι τρίτε χώρε, όπου να έχουμε κέρδο από τι παραγωγέ, λόγω χάρη με τη Ρουμανία, μια χώρα που θα μπορούσε λόγω χάρη να βοηθήσει να μειώσουμε, όχι να μηδενίσουμε, αλλά τουλάχιστον να μειώσουμε την εξάρτησή μα από την Αμερικανική Ήπειρο σε σχέση τουλάχιστον με την παραγωγή πρωτεϊνών ε, φυτικών. Κατά την άποψή σα, τι στρατηγική θα έπρεπε να χαράξουμε σε επίπεδο ΚΑΠ κυρίω και όπω είπατε κι εσεί, οι θετικέ πρωτενε έχουν αποτελέσει αντικείμενο αποσυνδεδεμένων βοηθειών, μάλλον συγγνώμη, συνδεδεμένων βοηθειών. Και θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα ποσοστό ώστε να ευνοηθεί η καλλιεργιά του, αλλά από την άλλη να προβλέψουμε λίγο και το μέλλον. Κατά την άποψή σα, λοιπόν, ποια στρατηγική πρέπει να θεσπίσουμε για να γίνει ευρωπαϊκή αυτή η προσέγγιση και να, μειώσουμε την, να περιορίσουμε την εξάρτησή μας. Ιδίω ως προς τις χώρες εντός της Ευρώπης. Να, να αναφέρω, θα μπορούσα να αναφέρω δύο, αλλά έχουμε και τις γείτονες χώρες όπως Ουκρανία, Ρωσία. Δηλαδή να έχουμε χώρες γειτονιά μας με τις οποίες να συνεργαζόμαστε και κάπως καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Διάβασα εδώ την έκθεση 2011 του Κοινοβουλίου για τα Μα χρονίζουν τα προβλήματα του ελλείμματος σε πρωτεϊνούχα. Την γνωρίζω καλά, άλλωστε γιατί ήμουν και συντάκτης. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο κενό έλλειμμα δεν αντιμετωπίζεται και ε, ε, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι τα υπολογίζουμε όλα ως μέτρα greening. Δεν φέρνουν αποτέλεσμα όμως. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ισχυρά γκλόμπι που δεν έχουν κανένα συμφέρον οι Ευρωπαίοι να παράγουν το δικό τους, τη δική τους πρωτεΐνη. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό λίγο καλύτερα. Αναφέρθηκε και η συμφωνία Blair House. Μήπως πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα και από πολιτική σκοπιάς. Έκανα νωρίτερα μια σύγκριση της παραγωγής μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, γιατί η παραγωγή της σόγιας στη Βραζιλία, όπως και στην Αργεντινή εξάλλου, δεν είναι αηφόρο, είναι πάρα πολύ εντατική δεν μπορεί να είναι η φόρα και γι' αυτό ερωτώ. Γιατί δεν έχουμε προχωρήσει, γιατί δεν έχουμε ενσωματώσει στόχους κλιματικής προστασίας, ε, προσδιορισμό επιβάρυνσης ε, στην περίπτωση παραγωγής ε, οξυδίων του αζότου, έτσι ώστε να συνδεθούν με την τιμή. Ο Ενεργειακός Επίτροπος έχει πει επίσης ότι πρέπει τα μέτρα που θα έχουμε στην παραγωγή πρωτενιούχων να συμβάλλουν περισσότερο, αλλά τα έχουμε επί χάρτου, δεν έχουν υλοποιηθεί διάφορα μέτρα. Το τριφύλι. Μηδική Δεν το αναφέρατε. Νομίζω ότι μπορεί και αυτό να... Αλλά δεν ε, αρκούν τα μέτρα αυτά. Οι βιολογικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι μπορούμε και χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Γιατί δεν προχωρούμε προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν. Πάνω απ' όλα λοιπόν το έλλειμμα για μένα είναι ότι υπάρχει έλλειμμα ε, γνώσεως στην παραδοσιακή ή συμβατική θα λέγαμε καλύτερα η ε, καλλιέργεια και γεωργία. Δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα με την καλλιέργεια ε, τα κτλ. Ναι, να σας πω εγώ το, στο θέμα αυτό ε, μυδικής κτλ. δεν ε, επεκτάθηκα γιατί δεν ήταν στο θέμα μου ακριβώς, αλλά το Σάββατο ήμουνα σε μια εκμετάλλευση που γνωρίζω εδώ και χρόνια. Το πρόβλημα που έχει είναι ότι ε, δεν μπορεί να έχει ποσοστό άνω του 1 τρίτου των εσόδων της από ε, τις ε, βιολογικές καλλιέργειες. Πρέπει να εξαρτάται οπωσδήποτε από τη συμβατική καλλιέργεια. Και βεβαίως έχετε δίκαιο ότι έχουν κάνει πολλά στον τομέα οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις, αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι μερικές φορές έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και έτσι αυτό είτε ε, όταν θέλουμε να αλλάξουμε, ε, ε, πρέπει να εξεταστεί όταν θέλουμε να αλλάξουμε από, το, από τη συμβατική καλλιέργεια ή αν θέλουμε να επεκτείνουμε τη βιολογική. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και με εκμεταλλεύσεις βιολογικής καλλιέργειας επαφή και συνεργασία αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τη βιολογική γεωργία. Ένα ζήτημα το οποίο έχουμε παραδείγματι αγνοήσει ότι δεν έχουμε κάνει αρκετή έρευνα δηλαδή και δεν έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα αυτά και αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα πρωτεϊνούχα δεν καλλιεργούνται κιόλας. Έχουμε λοιπόν ένα φαύλο κύκλο που πρέπει να σπάσουμε αυτή τη στιγμή. Εάν μπορέσουμε με κίνητρα, κυρίω με κίνητρα όπω ε, αυτό του πρασινίσματο που αναφέραμε νωρίτερα, μπορούμε να περάσουμε σε μια ε, εξέλιξη καλλιέργεια που θα έχει και την αηφορία μαζί. Σα ευχαριστώ. Κύριο Άλφερντ, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας. Πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν μπορώ να τα υποστηρίξω. Εγώ είχα κάνει ε, καλλιέργειες από πολύ νωρίς σε ε, ψυχανθή και μπόρεσα και με χειμερινή ε, καλλιέργεια να έχω καλή απόδοση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υποστήριξη από τους ε, τεχνικούς, από τους επιστήμονες και νομίζω ότι Ε, σε σχέση με το παράδειγμα της Βραζιλίας, αγαπητέ κυρία Χόισλινγκ που αναφέρατε νωρίτερα, υπάρχουν ε, τεράστιες καλλιέργειες. Ε, εγώ γνωρίζω γεωκτήμονα με 2.400 εκτάρια που όμως μπορούν να έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση και με σωστή εναλλαγή στη σπορά να διατηρούν την παραγωγικότητα, τη γονιμότητά τους. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορούμε να κοιτάξουμε είναι το πώς ε, ε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και τα μηχανήματα για την παραγωγή και τις ε, και των ε, ψυχανθών βεβαίως για την ε, ε, ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για ζωοτροφές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το είδαμε και στη χθεσινή συνεδρίαση, είναι να προχωρήσει με κατεξουσιοδότηση πράξης, τις οποίες όμως θα πρέπει, εάν επιμείνει στις ε, επιλογές της η Επιτροπή, να απορρίψουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα διαπραγμάτευση, κύριε Χόισλινγκ. Εγώ νομίζω ότι ήταν ε, σχεδόν ομόφωνη η απόφαση που λάβαμε εδώ στην Επιτροπή για να προτείνουμε την υποστήριξη των καλλιεργειών αυτών, των πρωτεϊνούχων, ώστε να σταματήσουμε να εξαρτώμεθα από τις, εξαγωγές, από τις εισαγωγές. Ευχαριστώ. Λουαζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως το ξέρουμε καλά εδώ, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την εκτροφή των ζώων σε τροφές πλούσιες αμινοξέα και πρωτεΐνες. Όμω, όσα ήδη καλλιεργούνται στην Ευρώπη δεν καλύπτουν παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό των ε, αναγκών των εκμεταλλεύσεων και τη κοινοτροφία. Για την, για την ελαιοκράμπη λόγου χάρη και τη σόγια είναι μόνο το 24%. Η Γαλλία και η Ευρώπη εισάγουν ε, πολύ, μεγάλα, πολύ μεγάλου όγκου από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη ΣΥΠΑ και η σόγια σήμερα είναι η θύρα που θα επιτρέψει την είσοδο των γάμα ταφ στην Ευρώπη, των γάμα ταφ όμικρων που προκαλούνται και υποψία των καταναλωτών, όπω ξέρετε καλά. Αυτή λοιπόν η εξάρτηση, διότι είμαστε προ τη αγωγή και καταναλωτέ ε, αυτών των προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανική επεξεργασία ελαίων, και επειδή όλα αυτά διέπονται και από συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, όπω με τη Λευκορωσία, με τη Ρωσία μάλλον το 1992, αλλά και την Ευρώπη και τις ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε πως έχει διαμορφωθεί η επιφάνεια καλλιέργειας ελόγων πρωτεϊνών στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Ειδικά στη Γαλλία θέλουμε τη σχετική εξάρτηση από την εισαγωγή σόγιας να την περιορίσουμε, γιατί ακριβώς αυτή η σόγια είναι κυρίως γενετικώς τροποποιημένη. Η Γαλλία έχει δυναμικό για 200.000 εκτάρια βάσει των επαγγελματίων του χώρου, και θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τις 100.000 εκτάρια που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή με 40.000 εκτάρια 140 να, έχουν ήδη χρησιμο... να χρησιμοποιούνται ήδη το 2014. Ένα πολύ μεγάλο μέρο λοιπόν των πρωτεϊνών μα στη Γαλλία εισάγονται. Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε την καλλιέργεια όλων αυτών που μα λείπουν για να φτάσουμε στην αυτάρκεια. Τι προτείνετε εσεί για να δώσουμε κίνητρα με τρόπο συγκεκριμένο και χειροπιαστό στη οι να αυξήσουν την επιφάνεια παραγωγή των ελόχων πρωτεϊνών, ιδίω τη όγια. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να έχουμε κτηνοτροφία χωρίς να έχουμε και την κατάλληλη, τις κατάλληλες ζωοτροφές. Βεβαίω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εκπομπέ αερίου του, θερμοκηπίου, του του μεθανίου. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τόσο, τόσο μεγάλε εισαγωγέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί στου φυσικού πόρου, και είναι πολλά τα κρατημέλη που δεν καλλιεργούν αρκετή σόγια. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Αλλά θα πρέπει, συνάδελφοι, να είμαστε ακριβοδίκαιοι όταν κάνουμε αυτό το είδου την ανάλυση. Διότι πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουν τόσε εισαγωγέ από τη Βραζιλία. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη αρκετέ ε, ποσότητε σόγια. Ακριβώ γιατί ανατώνω είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο κόστο. Αυτά που εισάγουμε από τη Βραζιλία είναι φτηνά εισάγουμε προϊόντα γενετικώς τροποποιημένης σόγιας και κανείς δεν μπορεί να μου να αντικρούσει αυτό το επιχειρήμα, αυτή τη διαπίστωση, αλλά πρέπει να δούμε γιατί λέμε όχι στην ε, δυνατότητα, την πιθανότητα καλλιέργειας της σόγιας εντό Ευρώπη την οποία έτσι κι αλλιώ καταναλώνουμε. Ε, σε αυτή την κατάσταση έχουμε φτάσει. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν έχετε εξετάσει το κόστος. Το κόστος που θα υπήρχε ανατόνου όταν παράγεται στην Βραζιλία από τη μία και από την άλλη σε αντιδιαστολή με τον ίδιο τόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε τις ε, διαφορές, διότι ποιος ασχολείται με τη Γεωργία γνωρίζει πολύ καλά ότι για ένα εκτάριο για την καλλιέργεια της ε, γενετικώς τροπημένης σόγιας υπάρχει ένας τρόπος, μία μονοτεχνική. Ενώ για την παραδοσιακή σόγια χρειάζονται πάρα πολλές φορές. Άρα εξηγείται και διαφορά στο κόστο. Εάν θέλουμε όμω να είμαστε ακριβεί, πρέπει να δούμε τι ακριβώ κάνουμε κιόλα. Δηλαδή, συμφωνώ να προωθήσουμε τι ελαιούχε ζωοτρεφέ και με γενετικώ τροποποιημένα συστατικά. Όμω πρέπει να βρούμε όλου του απαραίτητου πόρου, πολιτικού, τελωνιακού και το καθεξής εάν δεν θέλουμε τις ζωοτροφές που να είναι γενετικώ τροποποιημένες στα συστατικά του. Και πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδαλώ θα αναπαράγουμε στο δίνακε αυτό που ήδη συμβαίνει. ξεχνώντα το σημαντικότερο. Δηλαδή την τιμή της ζωοτροφής ανατόνω. Ευχαριστώ Ακούσαμε τους ομιλητές μας εδώ για πολύ διαφορετικά θέματα, τα οποία όλα καταλήγουν στο θέμα του πώς θα ε, ταΐσουμε τον κόσμο. Ακούσαμε και υπουργούς Γεωργίας εδώ, μας λέγανε ότι θα ταΐσουν τον κόσμο και ο Αμερικανός υπουργό μας είπε το ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ταΐσουν τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι έχει ένα πλάνο για να θρέψει τον κόσμο, για, την, ε, για τον παγκόσμιο πληθυσμό που θα αυξηθεί και ούτω καθεξής. Γιατί τι δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που να ταΐζουμε τους αυτούς μας, να θραφούμε μόνοι μας. Να τραφούμε μόνοι μας. Αυτό θα είχε μια λογική. Τι γίνεται με τον Βραζιλιάνο Υπουργό και τον Αμερικανό ε, Υπουργό που χέρι-χέρι θα πάνε στον ίδιο δρόμο να ταΐσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, με τι ε, κόστος υπάρχει κανένα συντονισμό για όλα αυτά ή το νόημα μήπως δεν είναι ακριβώς να τραφεί ο κόσμος. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει για να πάει και να προβλέψει Πώ θα φάει ο κόσμο που τον λυπάται. Θα έπρεπε ίσω, αλλά δεν το πιστεύω. Ε, νομίζω ότι όλο το θέμα είναι η απληστία, η αύξηση τη παραγωγή και η προσπάθεια να προσπαθείτε να ε, δημιουργήσετε περισσότερα προβλήματα στου ε, μικρούς γεωργούς, στους επιμέρους γεωργούς. Από πού προέκυψε λοιπόν αυτή η ιδέα ότι οφείλουμε να θρέψουμε τον κόσμο. Ε, διέπει όλα τα θέματα που συζητάμε εδώ και πραγματικά ειλικρινά ε, αρχίζω να αναρωτιέμαι για την εντυμότητα αυτής της ε, δήλωσης και της πρόθεσης. Ο κύριος Ανδριέ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους δύο εμπειρογνώμονες, τους δύο καθηγητές που μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ε, μελετών και ερευνών τους για το θέμα αυτό. Και να πω ότι ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι ε, θα μπορούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπνευστούμε, όπως είπε και ο κύριος ε, Ταραμπέλα, από την ιδέα να έχουμε ένα πραγματικά στρατηγικό σχέδιο για την ε, προμήθεια και τον ανεφοδιασμό μας σε φυτικές πρωτεΐνες στην Ευρώπη. Μας λείπει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο. Θα πρέπει όμως να συνδυάσουμε και να συντονίσουμε πολλές πολιτικές για να καταρτήσουμε ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο. Και σίγουρα η κοινή γεωρική πολιτική είναι αυτή που θα πρέπει να πρωτοστατήσει αυτή την προσπάθεια και είδαμε ότι είχαμε προβλήματα με τη σύνδεση στο να προσθέσουμε το 2% για να βοηθήσουμε τους γεωργούς μας να εξασφαλίσουν πρωτεϊνική αυτάρκεια. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να παρέμβει στο θέμα αυτό για να εξασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό μας σε θετικές πρωτεΐνες. Επίσης, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και την εμπορική μας πολιτική. Γιατί γνωρίζουμε ότι ε, δεν είναι πια επίκαιρη, είναι παροχημένη. Θα πρέπει να την προσαρμόσουμε ε, στην περιβαλλοντική μας πολιτική και στην ε, πολιτική της αναχέτησης και του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε τι συμβαίνει στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ όταν μαζικά εισάγουμε και τι γίνεται με την ε, ανάπτυξη των επιφανειών καλλιέργειας όγιας και πόσο αυτή γίνεται εις βάρος ε, του δάσους της Αμαζονίας ε, και πόσο έχουν αποψηλωθεί δασικές εκτάσεις ε, τροπικών και παρθένων δασών για να επεκταθούν οι εκτάσεις καλλιέργειας σόγιας. Προτάθηκε η Ουκρανία και η ιδέα να στραφούμε προς τους γείτονές μας. Νομίζω ότι με γειτονικέ χώρες θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε πολύ πιο θετικά και ευνοϊκά για μας. Επίσης, ε, είναι πολιτική μας ευθύνη να αναπτύξουμε και να εξασφαλίσουμε τα εφόδια και τα μέσα για την έρευνα. Γιατί στο θέμα αυτό θα πρέπει να συντονίσουμε τους μηχανισμούς και τα μέσα που έχουμε για να ανακτήσουμε μία ε, διατροφική αυτάρκεια. Δεν μιλούμε για να θρέψουμε ολόκληρο τον πλανήτη. Ας καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο βαθμό διατροφικής αυτάρκεια σε φυτική πρωτεΐνη και αυτό αρκεί. Ο κύριος Δεκάστρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτησή μου εν μέρη καλύφθηκε από τον συνάδελφο Μπούντα. Η Ευρώπη είναι σαφώς εισαγωγέας μεγάλων ποσοτήτων σόγιας από χώρες της Βορείου και Νοτιού Αμερικής, Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα αριθμό πραγματικά τεράστιος, εκατοντάδες ε, χιλιάδων τόνων. Θέλαμε με την ΚΑΠ να δώσουμε περισσότερα κίνητρα ώστε η ευρωπαϊκή παραγωγή σόγιας να αυξηθεί και να βελτιωθεί. Αυτό δεν αλλάζει το ότι οι αυξήσει που υπάρχουν, οι μελέτες σας το επιβεβαιώνουν, είναι ακόμα πολύ σχετικές. Η ερώτησή μου λοιπόν επαναλαμβάνει λίγο αυτή του κυρίου Μπούντα προηγουμένω. Μπορούμε να καταφέρουμε αύξηση τη παραγωγή ελαιόχων πρωτεϊνών στην Ευρώπη, λαμβάνοντα υπόψη ότι 19 από τι 28 χώρε έχουν απαγορεύσει την καλλιέργεια ελαιούχων πρωτεϊνών και γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στο εδαφός τους. Υπάρχει πραγματική δυνατότητα να μεγαλώνουν τα φυτά ελαιούχων πρωτεϊνών στην Ευρώπη χωρίς χρήση γενετικώ τροποποιημένων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ μόν δεν θέλει να τα καλλιεργεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μας ανέφεραν οι ομιλητές μας τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα των εισαγωγών σόγιας. Θα μας εξηγήσετε τι εννοείται ως αποδεκτά επίπεδα εισαγωγών. Γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ ψηλό το 70% που εισάγουμε, αλλά ρεαλιστικό τι θα ήταν, τι θα ήταν ε, πιθανό να μπορούμε να υποκαταστήσουμε ως παραγωγή από την εισαγόμενη. Και επίσης μη γενετικά τροποποιημένη σόγια είναι ρεαλιστικό να καλλιεργήσει ο Ευρωπαίος Γεωργός. Τρίτον, οι δασμοί εισαγωγικοί. Τι συνέπειες μπορούν να έχουν στο κόστος και την παραγωγή τροφίμων. Εάν τυχόν και αποφασίσουμε μια σκληρή πολιτική να επιβάλλουμε δασμούς για να ενθαρρύνουμε την εσωτερική παραγωγή. Τι συνέπειες θα είχε αυτό. Ευχαριστώ, Ντενανού. Πρόεδρε, ευχαριστώ ως ε, περιφερειάρχης προσπαθούσα να πείσω τους ε, καλλιεργητές και τους κτηνοτρόφους να καλλιεργούν οι ίδιοι πρωτεϊνούχα φυτά στις εκτάσεις τους. Πολύ δύσκολο όμως ήταν αυτό, δεν ήταν εύκολο να τους πείσω. Ε, πότε μου λέγανε ότι δεν είχαν κατάλληλο χώμα, έδαφος ή ότι δεν είχαν αρκετό νερό ή ότι είχαν παραπάνω νερό ή ότι είχαν ε, ανεπαρκή κατάρτιση για την ε, καλλιέργεια. Εν πάση περιπτώσει, τι είδους εργαλεία πρέπει να διαθέσουμε σε αυτούς τους καλλιεργητές για να τους επιτρέψουμε μέσα στην εκμεταλλεύση τους τα εδάφη τους να προωθήσουν την καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων, γιατί έτσι νομίζω σε ένα στενό στον εγκύτερο δηλαδή, στην εγκύτερη περιοχή γεωγραφικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτές τις καλλιεργίες. Και ο κύριος, Χόισλινγκ ξαναζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, αλλά να είστε σύντομος. Ναι, πολύ σύντομα, διότι το πρόβλημα που είχαμε στην ε, συζήτηση ήταν και το επιβεβαίωσε ο κύριος Δες ότι η Ευρωπαίοι παραγωγοί καλλιεργητές και φτώνταν μόνο κόλζα όταν γινόταν λόγος για πρωτεϊνούχα που ούτως ή ε, δεν είναι καν, είναι ελαιούχο φυτό περισσότερο. Ε, για τα ψυχανθή δεν γινόταν αρκετός ε, λόγος και μάλιστα πάνω απ' όλα δεν γινόταν λόγος για το ότι μπορεί να βοηθήσει και στον περιορισμό των ε, ποσοστών, ε, των ποσοτήτων ε, οξυδίων του αζότου που ανοιχνεύονται στην ατμόσφαιρα. Έχει μεγάλο δυναμικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε μπορέσει και στη δική μου την περιοχή να κάνουμε καλλιέργειες. Γιατί να μην καλλιεργούμε λοιπόν ευρωπαϊκή σόγια ή να ανοίξουμε τη συζήτηση και να δούμε τι άλλα υποκατάστατα μπορεί να υπάρχουν. Και γνωρίζω ότι μπορεί κανείς να έχει ένα παράδειγμα με τον περίφημο βραζιλιάνο γεωκτήμονα που έχει αηφόρο παραγωγή κτλ. Αλλά δεν μπορεί με ένα παράδειγμα να αγνοούμε ή να, να αρνούμε θα την πραγματικότητα. Έχουν ε, πολύ εντατική καλλιέργεια στην ε, Αμερική, στην Αργεντινή και τη Βραζιλία συγκεκριμένα ε, και σε πράγματα στα οποία εμείς, σε παραγωγές στις οποίες εμείς δεν έχουμε αρκετές, ε, αρκετούς όγκους, αρκετές ποσότητες, εκείνοι μπορεί να έχουν υπερβολικές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και πάλι στους καλεσμένους μας. Α, συγγνώμη. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευχαριστώ τους καλεσμένους σας ε, για τις παρουσιάσεις που έκαναν και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, λίγα σχόλια θα κάνω μόνο. Ε, αυτό που φάνηκε και από τις παρουσιάσεις και από τη συζήτηση είναι οι οικονομικοί παράγοντες ε, που οδηγούν τους γεωργούς να μην επιλέγουν τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Επίσης, να αποσαφηρήσουμε και το εμπορικό καθεστώς. Όντως, οι ελαιούχοι σπόροι και ε, οι πρωτεϊνούχες πόλοι έχουν ε, ελάχιστους ε, δασμούς ή μηδενικούς, αλλά το ίδιο ισχύει και για τα σιτηρά, τα δημητριακά, και εντός και εκτός των συνόρων. Οπότε οι ίδιες αθασμολόγια της εισαγωγές ισχύουν και για άλλα προϊόντα. Τώρα για την κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος μέσων και εργαλείων που έχουμε αυτή τη στιγμή για να ξεπεράσουμε τους στενούς οικονομικούς παράγοντες και σίγουρα ε, έχουμε με τις άμεσες ενισχύσεις ε, ένα, μια προστασία του εισοδήματος και το πρασίνισμα επίσης λαμβάνεται υπόψη για τα περιβαλλοντικά ωφέλη Επίσης στο πρασίνισμα έχουμε και την απέτηση για, τις, για τους χώρους οικολογικής εστίασης και το θέμα της αμύψης ποράς είναι πολύ σημαντικό. Με την αμύψης πορά δίνουμε κίνητρα ε, για καλλιέργειες και πρωτεϊνούχων φυτών. Και οι επιλογές των κρατών μελών επίσης είναι σημαντικές. Ε, η αγροτική ανάπτυξη, ανάπτυξη πέθρου για πολλά χρόνια παρέχει στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Κάποιος ανέφερε κάποια στοιχεία για την έρευνα και τα κονδύλια που αφιερώνονται στην έρευνα για το θέμα αυτό. Στο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7, αλλά και στο Erasmus ε, και στο Ευρώπη 2020, ε, έχουμε κάποια ερευνητικά προγράμματα πανευρωπαϊκά, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα της έρευνας γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Καινοτομία έχει μια ειδική ομάδα που επικεντρώνεται στα πρωτεϊνούχα φυτά. Και βλέπουμε μια αντιστροφή αυτής της τάσης. Κάποιες εξελίξεις και βλέπουμε ότι ο οικονομικός παράγον δεν είναι ο μόνος που λαμβάνεται πια υπόψη. Ούτε η κατάσταση είναι μονοσήμαντη. Γιατί στις ε, γεωργικές πρακτικές των Ευρωπαίων Γεωργών αλλά και στην αμυψησπορά οι, τα πρωτεϊνούχα φυτά, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες αρχίζουν και παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο και αυτή την ναι. τάση θα προσπαθήσουμε να την ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Κύριε καθηγητά, πέντε λεπτό καθένας παρακαλώ. Το πολύ. Ja, es waren eine ganze Reihe von... Ναι, μια σειρά από που με αφορούν. Θα συνεχίσω αυτό που είπε ο κύριος Χόισλινγκ. Με συγχωρείτε κάτι. Ξέχασα, ξέχασα τι με ρωτούσατε. Θα μου το θυμίσετε κύριε Χόισλινγκ. Πολύ σύντομα. Αυτό με την αντικατάσταση ευρωπαϊκής σόγιας από εισαγω... της από ευρωπαϊκή αλλά και άλλες εναλλακτικέ καλλιέργειες. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ, ότι έχουμε πολλέ πολλές ε, ενδιαφέρουσες καλλιέργειες και στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουμε σημαντικές ε, τέτοιες παραγωγές που ε, καλύπτουν τις ανάγκες ε, σε σόγια σε ένα μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν περιορισμοί στην Ευρώπη που έχουν να κάνουν με την ε, εναλλαγή των καλλιεργειών και ακριβώς εκεί είναι οι περιορισμοί. Εάν λοιπόν θέλουμε να ε, δούμε το ποσοστό για τα ψυχανθή, ε, είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα να τα αντικαταστήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή πλήρως να αντικαταστήσουμε τη σόγια από μια άλλη καλλιέργεια. Λόγω των περιορισμών στις ε, εναλλαγέ των καλλιεργειών, στη Γερμανία τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καν δυνατόν. Κύριε καθηγητά Γκονσόφσκι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι σε ό,τι αφορά τις αναλύσεις που έγιναν, έλαβε υπόψη μια έκθεση για, για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πρωτεϊν, πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως, ήταν η βάση για την ανάλυση και αναφέρει και τους, τις μεθόδους επίλυσης του προβλήματος. Δεν ήθελα να επαναλάβω ότι έχουμε ε, υπερπαραγωγή στα δημητριακά. Είμαστε ο πρώτος εξαγωγέας δημητριακών στην Ευρώπη, κυρίως σε ΣΥΤΟΥ. Σε, αντίθεση με το ΣΥΤΟΥ όμως που είμαστε με ο πρώτος εξαγωγέας, είμαστε πολύ σημαντικός εξαγωγέας σόγιας, δεύτερος παγκοσμίως. Αυτή τη διαφορά, αυτή την ισορροπία θα πρέπει να την διορθώσουμε. Το είπαν και οι ευρωβουλευτές. Σε ό,τι αφορά ε, τα άλλα ψυχανθή και τις μερικές φορές οι, οι αποδόσεις ε, των ε, καλλιεργιών δεν είναι ίσες. Θα πρέπει για να διορθώσουμε την κατάσταση να λάβουμε υπόψη τον οικονομικό παράγοντα και να κάνουμε πιο οικονομικά ελκυστικέ τις καλλιέργειε ψυχανθών. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή των τροφίμων έχουμε μια τεχνητή πλασματική κατάσταση και όπως είπαν οι Υπουργοί Γεωργίας ε, της ε, Βραζιλίας και των Ηνωμένων Πολιτικών, ε, θέλουμε, είπαμε, να, είπαν να θρέψουμε όλο τον κόσμο, αλλά τι γίνεται στην υποσαχάριο Αφρική. Σήμερα είναι 800.000 άνθρωποι, σε λίγους δεκαετίες θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Ήδη υπάρχει πρόβλημα υποσυτισμού και ήδη υπάρχει έλλειμμα στην παραγωγή τροφίμων στην υποσαχάριο Αφρική όσο περισσότερο αυξάνονται τα προβλήματα και οι δημογραφικές πιέσεις, θα έχουμε μία έξοδο μεταναστευτική από την υποσαχάρια Αφρική προς την ε, Ευρώπη με τις ε, αναμενόμενες συνέπειες. Επίσης, ε, εγώ πρότεινα να επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές πρωτεϊνοχων φυτών. Βέβαια αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε. Ε, δεν το ανέφερε ο πρόεδρος, αλλά εγώ ξεκίνησα ως ε, γεωργός και ασχολήθηκα μια δεκαετία με το θέμα αυτό και με την καλλιέργεια σιτηρών. Και νομίζω ότι ακόμη και τώρα να ξεκινήσουμε πιο εκτεταμένη παραγωγή ψυχανθών θα χρειαστούμε 5 με 10 χρόνια για να έχουμε μια υψηλότερη απόδοση των καλλιεργιών αυτών. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον παράγοντα χρόνο. Επίσης, ε, ε, να μην ξεχνούμε ότι Εκτός από τη σόγια έχουμε και άλλα ψυχανθή που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή πρωτεϊνών αντικαθιστώντας τη σόγια. Δεν είναι μόνο η σόγια ψυχανθές, υπάρχουν και άλλα πρωτεϊνούχα φυτά. Επίσης, ε, από ό,τι ξέρω, χωρίς απόφαση με οικονομικό χαρακτήρα, και εδώ αναφέρθηκε το θέμα των επιλογών της ε, γεωργικής πολιτικής στη Βραζιλία, θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι όταν υιοθετήθηκε η κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώθηκε η επιφάνεια καλλιέργειας ψυχανθών, ενώ αυξήθηκε η καλλιέργηση επιφάνεια δημητριακών και κυρίως σύτου, ενώ προηγουμένως είχαμε την αντίθετη κατάσταση. Οπότε δεν είναι μόνο οικονομικές οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν, αλλά πρώτα απ' όλα πολιτικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ολοκληρώνουμε το πρώτο τμήμα της δημόσιας ακρόασης μας και περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ματίας Κχέν. κατόπιν η κυρία Μαρία Πελετιέ, και τέλος ο κύριος Ντέιβιτ Μακνότον. Ο κύριος Ματίας Κρόν θα μας μιλήσει για την ε, διαφοροποίηση των ε, καλλιεργειών ψυχανθών και το ρόλο της όγιας στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία καθώς και την Ευρωπαϊκή Μετάβαση σε πρωτεΐνες. Ο κύριος Κρέν είναι πρόεδρος της ε, Ένωσης Σόγιας του Δούναβη, που είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση ε, που ε, προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς μεταλλαγμένη σόγια παραγωγή κατά μήκο του Δούναβη από την Ελβετία μέχρι τον Ευξηνοπόντο. Παρακαλώ κύριε καθηγητά, κύριε Κρέν, έχετε το λόγο. Good afternoon. I hope you can all hear me. My name is Matthias Krohn. I'm very happy to be here. Okay. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Κάτι δεν πάει καλά με τις διαφάνειές μου, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχω μόνο μία διαφάνεια και δεν είναι πάρα πολύ σημαντική για την παρουσίαση μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω και τους δύο προλαλήσαντες, τον κύριο Κοσόφσκι και τον κύριο Σέφερ, έθιξαν πολλά θέματα που ήθελα και εγώ να καλύψω με τη σύντομη μιλία μου. Όπως προβλέπει το πρόγραμμά σας για σήμερα, ήθελα να μιλήσω για το ρόλο της όγιας στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, βασιζόμενος στην ε, επίρα που έχουμε στην πράξη από τον οργανισμό Σόγια του Δούναβη. Μια διεθνή με κυβερνητική οργάνωση με 245 μέλη σε 19 ευρωπαϊκές χώρες. Η έδρα μας είναι στη Βιέννη. Δεν είμαστε λόμπι της Σόγιας, δεν έχουμε οικονομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε, είμαστε μια πρωτοβουλία της περιοχής του Δούναβη και έχουμε μέλη παραγωγών ε, γεωργικών συνεταιριστικών, εταιριών επεξεργασίας τροφίμων, ε, κτηνοτροφίας, γενοπολιτών, ενώσεων των πολιτών και ούτω καθεξής. Είμαστε μια μεγάλη οργάνωση. Μιλάμε για τη σόγια στην περιοχή μας, γιατί είμαστε από την περιοχή του Δούναβη και είναι το ψυχανθές που καλύτερα έχει προσαρμοστεί στη δική μας την περιοχή και μάλιστα από πολύ καιρό, 150 χρόνια τώρα. Περισσότερο από ότι οι Αμερικανοί, οι Βραζιλιάνοι ή οποιοδήποτε άλλος εκτός από τους Κινέζους και τους Ιαπωνέζους. Η σόγια λοιπόν είναι ένα παραδοσιακό ευρωπαϊκό φυτό του Δούναβη και έχει ριζώσει σε εμά. Έχει όλα τα ωφέλη των άλλων ψυχανθών, ε, την ε, πολύ καλή προσαρμογή του στο έδαφο, είναι πολύ καλό για τι υπόλοιπε καλλιέργειε. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην συζητάμε τη σόγια εναντί τη σόγια, αλλά τη καλή και τη κακή γεωργική πρακτική. Των καλών συστημάτων ε, συγκομιδή και όχι. Θα ήθελα λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα από μια κάπω διαφορετική προοπτική. Διότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά φυτά, υπάρχουν καλά ή κακά συστήματα πιστεύω. Και εδώ μιλάμε για βελτίωση του γεωργικού μα συστήματο με τη σόγια στην περιοχή μα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η μόνη λύση. Υπάρχουν και άλλα καλά ψυχανθή σε άλλε περιοχέ παραγωγή. Λοιπόν, το ε, ζήτημα δεν είναι υπέρ κατά τα μείον και τα συν, αλλά το τι θέλουμε εμεί να πετύχουμε. Το θέμα μας όμως είναι διαφορετικό. Η πρωτεϊνούχα μετάβαση η μετάβαση στην πρωτεΐνη. Όπως με την ενεργειακή μετάβαση, μιλάμε για την αλλαγή της καλλιέργειας στα εδάφη προς τα ανανεώσιμα βιώσιμα καύσιμα από τα ορεκτά. Το ίδιο θέλουμε να συμβεί και με τι καλλιέργειε. Να σα εξηγήσω πώ το βλέπουμε λοιπόν αυτό και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε. Τι μα κινητοποιεί. Όπω είπα, θέλουμε καλύτερη και πιο ποικίλη ε, εναλλαγή των ε, καλλιεργειών παγκοσμίω. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Αν δείτε, τι γίνεται, αν δείτε στην Λατινική Αμερική, κατά μέσο όρο μέρο όλων των καλλιεργειών είναι το 77% στην Παραγουάη μόνο και το περίπου 60% στον κόσμο, ε, στο, στην Ήπειρο, στο έδαφος, Είναι υπερβολικά πολύ η σόγια της Λατίνική Αμερικής, δεν είναι υγιές και δεν είναι καλό για τη γεωργία, αλλά ούτε και βιώσιμο αυτό το σύστημα. Στην Ευρώπη έχουμε 2% ε, της αεροτρέας γης ε, με ψυχανθή και 0,9% σόγια. Δεν έχουμε αρκετά ψυχανθή σόγια στην Ευρώπη και δεν έχουμε και αρκετή σόγια. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα ψυχανθή. Όλοι νομίζω θα συμφωνήσουμε. Όπω προείπα, τα ψυχανθή από μόνα του δεν είναι καλά ή κακά. Μόνο αν τα συστήματα είναι καλά μπορούμε να τα πούμε καλά και τα φυτά. Αυτό είναι πραγματικά καθοριστικό για να καταλάβουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε να προωθήσουμε τη σόγια, αλλά τη βελτίωση των συστημάτων καλλιέργεια. Δηλαδή και περισσότερη ανθεκτικότητα στο σύστημα παραγωγή, αλλά και περισσότερη ανεξαρτησία από τι εξαγωγέ. Ήθελα να σα κάνω πέντε σύντομε παρατηρήσει. Πρώτον, Έχουμε ακούσει την συζήτηση βιολογικής έναντι συμβατική καλλιεργίας. Εγώ ως μέλος οργάνωσης που ε, θέλει περισσότερα ψυχανθεί, αλλά όχι μόνο για πολιτικά κίνητρα που πηγάζουν από τις Βρυξέλλες, ούτε από τους δύο καλλιεργητές, αλλά και από τους παραδοσιακούς γεωργούς η παραδοσιακή γεωργία τα ζητάνε όλο και περισσότερο. Μιλώντα λοιπόν από μια τέτοια οργάνωση, πρέπει να πω ότι αυτό χρειάζεται για να έχουμε περισσότερη συγκομιδή, περισσότερη σοβιά, να μειώσουμε τη χρήση ε, και φυτοκτόνων, για να μειώσουμε το κόστο παραγωγή ε, και τα προβλήματα ε, χρήση του εδάφου. Οι γεωργοί θέλουν ε, την χρήση τέτοιων συστημάτων για καλύτερες επιδόσεις. λόγω χάρη στην Αυστρία η σόγια είναι από τις καλύτερες καλλιέργειε τα τελευταία 10 χρόνια, από τις πιο ανταγωνιστικές. Το έδειξαν ανεξάρτητες μελέτες. Η σόγια λοιπόν και άλλα ψυχανθή μπορεί να είναι ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Εάν δούμε την τιμή για τα θέματα αυτά, παρατηρήσουμε ότι οι τιμέ στην Ευρώπη ε, υποφέρουν και πλήττονται από την υπεραπλούστευση. Ενώ θεωρητικά οι νέε ποικιλίε καλλιεργούνται περισσότερο, οι επιφάνειες που καλλιεργούνται δεν αυξάνονται, διότι τα συστήματα καλλιέργειά μας δεν είναι αρκετά ποικίλα. Πρέπει λοιπόν να ε, βελτιώσουμε τη χρήση του εδάφους για να έχουμε περισσότερη παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Αυτό το λέει ανεξάρτητη μελέτη. Είναι πολύ σημαντικό να το παρατηρήσουμε. Δεύτερη παρατήρηση για την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Για την ΚΑΠ. Τα έχετε ακούσει και στο παρελθόν. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν αναγνωρίσει τη σημασία τη ε, διαφοροποίηση των συστηματοκαλλιέργεια ε, στην ΚΑΠ με διάφορα συστήματα μέτρηση. Αυτή τη στιγμή η ΚΑΠ έχει και φυτά που παράγουν ε, ε, αζωτούχα σε περιοχές πρασινίσματος, αζωτούχα αέρια, αλλά υπάρχει και μία τάση ύφεσης της χρήσης των ψυχανθών. Πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγή ψυχανθών με τέτοια μέτρα που να έχουμε περισσότερη εναλλαγή καλλιεργιών με ψυχανθή στην Ευρώπη. Είναι επικίνδυνο να πούμε ότι θα καταργήσουμε τις περιοχές ε, πρασινίσματος και τα ψυχανθή δεν μπορούν να καλλιεργούνται εκεί και να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν είμαι κατά των ψυχανθών στις περιοχές πρασινίσματος, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω, σε άλλο επίπεδο, λόγω χάρη στην εναλλαγή των καλλιεργιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική των πρωτεϊνών, δηλαδή να μειώσουμε τις εισαγωγές και να βελτιώσουμε τα συστήματα καλλιέργειας. Κοιτάξαμε από την ε, σκοπιά των εισαγωγών τι μπορεί να είναι βιώσιμο. Ως εξαγωγής θα έπρεπε να εξάγουμε τρόφιμα, αλλά όχι να εισάγουμε σόγια. Αυτό το βρίσκω εσφαλμένο. Όμω ε, η εξάρτησή μα πρέπει να μειωθεί για να είμαστε μακροποθέσμα βιώσιμοι. 35 ισοδύναμα των εκατομμύρια τόνων ε, εισάγουμε ετησίω στην Ευρώπη, ε, ενώ παράγουμε μόνο 2,5. Αυτό είναι επικίνδυνο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ζω στην Βιέννη, πολύ κοντά στην Ουγγαρία. Και αν κοιτάξω προ Ανατολά, προ τη Ρουμανία και ακόμη πιο μακριά προ την Ουκρανία, έχουμε περίπου 100 εκτάρια γη σε αυτή την ε, ε, περιοχή. Και είναι πολύ έφορη αυτή η γη οι εξαγωγεί συμφωνούν ότι θα πρέπει στην ίδια περιοχή να παράγουμε 40% περισσότερο τα επόμενα 20 χρόνια. Έχουμε λοιπόν χώρο και για περισσότερα ψυχανθά και ψυχανθή και για περισσότερο σύτο και για περισσότερε καλλιέργειε. Δεν είναι το θέμα να ε, αντιπαραθέσουμε τη σόγια με κάτι άλλο, αντιπαραβάλλουμε τη σόγια με κάτι άλλο, αλλά να αυξήσουμε τι καλλιέργειε. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με αυτό το 40% επιπλέον. Ε, θα έχουμε κακά συστήματα καλλιέργειας με 2% ψυχανθή στην Ευρώπη ή θα έχουμε την ίδια και για περισσότερες πρωτεΐνες και καλύτερες γεωργικές πρακτικές στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό οι να γνωρίσουν ότι δεν μιλούμε για ένα θέμα μηδενικής αντιστάθμισης, δηλαδή αντί για τη σόγια κάτι άλλο ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε όλα να τα καλλιεργήσουμε ταυτόχρονα. Ένα παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσουμε 5% τη ερωτρέας γη στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη, μπορούμε να παράγουμε τη μισή σόγια που χρειάζεται όλη η Ευρώπη. Δεν μιλάμε λοιπόν για μικρού αριθμού, 5% τη γη είναι περίπου ήδη το όγκο σόγια που παράγουμε στην Αυστρία. Ήδη. 5% τη γη θα έδινε 12 ε, περίπου εκατομμύρια τόνου σόγιας. Μιλάμε για τεράστιες, τεράστιους αριθμούς, τεράστιους Δεν είναι ε, ψίχουλα αυτά. Οπότε δεν μιλάμε ούτε καν για μονοκαλλιέργειες. Με εναλλαγή των ε, καλλιεργειών, με καλέ γεωργικέ πρακτικέ, θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Υπάρχουν λοιπόν περισσότερε ευκαιρίε ακόμη και αν στραφούμε προ τη Ρωσία Επόμενη παρατήρηση. Πρέπει κάτι να κάνουμε για την ανάπτυξη τη υπαίθρου και την προσφορά θέσεων εργασία στι περιοχέ τη υπαίθρου. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε περιοχέ πλεονάσματο στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη που εξάγουν ε, πολύ κοκό στάρι, στάρι, αραβόσιτο και φύτο για άλευρο. Αυτά συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και βουλιά για κάποιον που θέλει να επεξεργαστεί τα προϊόντα σόγια λόγου χάρη ήδη. Δεν μπορεί να εξάγουμε μόνο πρώτε ύλε. Αυτό είναι σύστημα αποκαιοκρατικό. Αυτό το έμαθα στο σχολείο. Οι απικίε ε, εισάγουν τι πρώτε ύλε και μετά εισάγουν τα τελικά προϊόντα. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Παραγώντα περισσότερη σόγια θα μπορούσαμε να στηρίζουμε και τι ευρωπαϊκέ εταιρείε για να μετατρέψουν τη σόγια, να την επεξεργαστούν και να τη χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήδη συμβαίνει, διότι ήδη με τους όγκους σόγιας που έχουμε, την διπλασιάσαμε την παραγωγή της σόγιας στα τελευταία πέντε χρόνια, από, 5.000 εκτάρια, από 500.000 εκτάρια σε περίπου ένα εκατομμύριο, και αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε επενδύσεις στις διάφορες εταιρείες με δημιουργία θέσεων εργασία σε όλες τις χώρες γύρω από το Δούναβι. Είναι κάτι που συμβαίνει λοιπόν ήδη και μπορούν περισσότερο να γίνουν και στην Ανατολική και στην Κεντρική Ευρώπη με περισσότερες θέσεις εργασία, ιδίω εφόσον έχουμε και ανεργία στις περιοχές της Υπέθρου και κρίση. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό αυτές οι πολιτικές να φέρουν και περισσότερες δουλειές στην Ευρώπη. Η σόγια για την Ευρώπη λοιπόν δεν είναι καλή ή κακή όπως τα άλλα Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημά μας και να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτή την ανάγκη που υπάρχει για πρωτεΐνη με την ε, βελτίωση των καλλιεργιών στην Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε στην ε, σόγια του Δούναβη ως ιδιωτική πρωτοβουλία για του δημόσιου συμφέρον. Επιδιώκουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην Ευρώπη. Διότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα σε μεγάλο επίπεδο, σε μεγάλη κλίμακα, όχι μόνο από τη δική μα την οργάνωση, αλλά και με άλλα ψυχανθή. Πρέπει να ενισχύσουμε κατά άλλα ψυχανθή σε άλλε χώρε, σε άλλε περιοχέ και όλα αυτά μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική μεταμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η φιλοδοξία είναι να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σίγουρα, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την ε, καλύτερη αλλαγή των ε, καλλιεργειών με καλύτερες γεωργικές πρακτικές και την οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κρέν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαρία Πελετιέ, που είναι μεταξύ άλλων μέλος της Γαλλικής Επιτροπής ε, Βιολογικής Γεωργίας και Αντιπρόεδρος της μη κυβερνητική οργάνωσης «Οι μελλοντικές γενιές» ε, που δραστηριοποιείται σε θέματα υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μαρία Πελετιέ. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να προσφέρω τη μαρτυρία μου ως οικονομικός παράγων της μακροβιολογίας εδώ και 30 χρόνια περίπου σε επίπεδο της επιχείρησης που διευθύνω Έχουμε μία επί της ουσίας δουλειά για την βιολογική ε, γεωργία και κυρίως την κτηνοτροφία και προσέξαμε μετά από τις σημερινές παρεμβάσεις ότι αυτό λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία διότι έχουμε και την ε, το είναι να συνεργαζόμαστε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να σα παρουσιάσω την επιχείρησή μα για να καταλάβετε πώ λειτουργούμε σε επίπεδο ε, επιχειρήση Λειτουργούμε από το 1984 και είμαστε τυχεροί διότι ασχολούμαστε με τι ε, σιτοφόρε λεκάνες ε, και με την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών. Είμαστε μια εταιρεία ανεξάρτητη και έχουμε πολλές ε, δραστηριότητες όπως την αλευροπία ε, και αρτοπία, την διατροφή των ζώων, την γεωργική βιολογία, την συγκομιδή και αποθήκευση δηλαδή συλλέγουμε θα που έχουμε συγκεντρώσει ως πρώτες από τους γεωργούς και μετά κάνουμε επεξεργασία προϊόντων και παραγωγή. Μας ενδιαφέρει η διαρκής ποιοτική έρευνα με εταιρική σχέση μαζί με χιλιάδες καλλιεργητές και γεωργούς κτηνοτρόφους την λογική μιας γεωγραφικής εγκύτητας η συνολική μας λογική μας επιτρέπει και να κοιτάζουμε τι γίνεται με τις καλλιέργειες, μετά να παίρνουμε σε τοπικό επίπεδο την παραγωγή της, συγκομιδή από τους ίδιους τους γεωργούς και ε, για την ζωοτροφή, τη διατροφή των ζώων, μιας και είναι το θέμα της ημέρας, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με ένα εργοστάσιο που πολύ συχνά επεξεργάζεται βιολογικά προϊόντα και σε αντίθεση με άλλες μορφές κτηνοτροφίας δεν αντιτασσόμαστε καθόλου στον εφηγονισμό, αλλά κοιτάζουμε πώς να προχωρήσουμε και από περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης με σύγχρονα εργαλεία. Καινοτομία λοιπόν, παρακολούθηση των κτηνοτρόφων και υποστήριξή τους, με λύσεις σκόπιμες σε συνεργασία με τα δίκτυα που έχουμε δημιουργήσει. Κτηνοτρόφοι, εργαστήρια, εμπειρογνωμοσύνη για την διατύπωση, για την πολύ σημαντική και η διατύπωση όταν μιλάμε για διατροφή των ζώων. Η συνταγογραφία μάλλον. Συνεργαζόμαστε με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ζώων, γιατί μας απασχολούν τα πουλερικά μέχρι τα σαλεγκάρια και άλλα, ε, άλλες περιπτώσεις όπως κάποια έντομα. Σε αυτή την επί της ουσίας δουλειά ε, κοιτάζουμε πάντοτε ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία των ζώων και την σωματική τους ακαιρεότητα. Ε, επίσης, μας απασχολεί και το οικονομικό κέρδος. Πρέπει να σεβαστούμε και τις διατροφικές και σωματικές ανάγκες των ζώων με τις ζωοτροφές που προσφέρουμε, με πρώτες ύλες γεωργικές, δεν χρησιμοποιούμε χημικά και τεχνητά προϊόντα, με τις πρώτες ύλες που διαθέτουμε διότι φροντίζουμε πρώτε ύλε να μα είναι διαθέσιμε από τι ίδιε τι γεωργικέ καλλιέργειε που παρακολουθούμε εμεί και να είναι κατευθείαν από τη γη. Έτσι, ε, κοιτάζουμε και το συνολικό κόστο ώστε και οι γεωργοί κτηνοτρόφοι να μπορούν να κερδίζουν τη ζωή του, να βιοπορίζονται από τη δουλειά αυτή. Η τεχνική επίση διάσταση μας απασχολεί πολύ, διότι εδώ και 30 χρόνια παρακολουθούμε τι κάνουν οι γεωργοί με οικονομικά αποτελέσματα πραγματικά σημαντικά. Σε επίπεδο από την άλλη έχουμε ανάγκη από την ποικιλία και τι πρώτες ύλες στη γεωργία, διότι όπω έλεγα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε χημικά προϊόντα, οπότε κοιτάζουμε να υπάρχει ποικιλία στην παραγωγή μας. Σε επίπεδο δημητριακών θα δείτε ότι έχουμε πολύ σημαντικό αριθμό ε, καλλιεργιών, σπορών με μεγάλη διαφορετικότητα ε, και έχουμε πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αυτό δίνει στους γεωργούς τη δυνατότητα να έχουν τεχνικές επιλογές ε, για να έχουν και διαφορετική κερδοφορία. Ως προς τα πρωτεϊνούχα έχουμε τα ψυχανθή, τα όσπρια, τα λούπινα, τους σπόρους σόγιας, τα τσόφλια από τη σόγια. Και όταν μιλάμε για την φυτική τους φλοιουσόγειας και όταν μιλάμε για την ε, ε, διατροφή των ζώων φροντίζουμε και εδώ τα υποπροϊόντα της συνολικής ε, παραγωγής τροφίμων να αξιοποιούνται. Όλα αυτά τα υποπροϊόντα λοιπόν, τα παραπροϊόντα, χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την κτηνοτροφία. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά προϊόντα και εδώ. Σόγια, ε, ηλιοτρόπιο, λινάρι, κάναβης, σουσάμι, ελαιοκράμβη, φλοιός ε, ε, ραχίδων, αμύγδαλα και ούτω καθεξής. Εδώ προσπαθούμε να δίνουμε ποικιλία διατροφής στα ζώα με διαφοροποιημένα στοιχεία που αυτό να επηρεάσει και την χρήση. Δηλαδή ακόμη και αν μιλάμε για παραγωγή μικρών ποσοτήτων φροντίζουμε να τις αξιοποιούμε σωστά. Θα τις ενσωματώσουμε μερικές φορές κατά 3, 10%, κάποιες φορές κατά 1% στην ε, τελική μας επιλογή. Αλλά φροντίζουμε όλα τα προϊόντα να αξιοποιούνται στην, στο φάσμα όλη της αλυσίδας. Επίσης ε, και ε, οι φυτικές πρωτεΐνες όπως πρωτεΐνη γεωμήλων, η γλουτένες, αλλά και αραβόσιτου μας καλύπτουν κάποιες από τις ανάγκες μας. Κοιτάζουμε επίση τα φυσικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών, όπω την ενέργεια, την πρωτενη, τι ίνε και ούτω καθεξή. Επίση το κόστο και τέλο την διαθεσιμότητα με ε, την σύναψη ανάλογων συμβάσεων. Μια από τι φόρμουλε που χρησιμοποιούμε και έχω πάρει μία στην τύχη ε, είναι ε, μια, ένα, ενα μοντέλο για το πώ χρησιμοποιούμε τι πρώτε ύλε για να επιφέρουμε τη σωστή εξισορρόπηση με τα ανάλογα τεχνικά αποτελέσματα. Βλέπετε με την Λουζέρ δείχνει τι γίνεται και το πώς η περιεκτικότητα έχει σε πρωτεΐνη. Χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία βοηδών, πουλερικών, ε, και για τις ε, και σόρνηθες όταν θέλουμε κίτρινα αυγά ή με τεχνητά προϊόντα. Εάν προσθέσουμε έλεγε λουζέν λόγου χάρη με αραβόσιτο τελικά καταλήγουμε στο αποτέλεσμα αυγό που θέλουμε και το επηρεάζουμε. Είμαστε πάντοτε λοιπόν σε αυτή την αναζήτηση εξισυρώπησης τεχνικών ε, και φυσικών χαρακτηριστικών αλλά και σωστής διατροφής για τα ζώα για να είναι καλά και η κερδοφορία να είναι ανάλογη με τις ανάγκες των ε, κτηνοτρόφων μας. Ως προς τα τεχνικά αποτελέσματα, τα τεχνικά αποτελέσματα τα παρακολουθούμε με εκθέσεις που γίνονται από τους ε, υπευθύνους μας, ε, γεωπόνους και ε, κτηνιατρούς, ιδίω για τα πολυερικά λόγω οτό και σόρνηθες, έχουμε αποτέλεσμα ανάλογο με τη συμβατική κτηνοτροφία με πολύ λιγότερη ανάγκη συμμετοχής και παρέμβασης κτηνιάτρου. Διότι διευθετούμε έτσι τη διατροφή που η παρέμβαση κτηνιάτρου δεν χρειάζεται τόσο, Ιδίω προς τη χρήση χημικών προϊόντων, είτε είναι ιατρικά προϊόντα, σκευάσματα είτε όχι. Η διατροφή που δίνουμε στα ζώα επιτρέπει ακριβώς αυτά τα ζώα να είναι σε καλή υγεία και η κερδοφορία μας να είναι και η σωστή. Δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν αυξητικά στοιχεία με τα λούπινα, τα άλλα όσπρια και... Ε, την ειδική πολλές και με, τα, με τις πίτες ηλιοτροπίων πολλές φορές καλύπτουμε τις ανάγκες ε, των ζώων σε πρωτεΐνες με πολύ σωστά ποσοστά και καταλήγουμε σε αποτέλεσματα πανομοιότυπα με τη συμβατική εκτενοτροφία χωρίς την χρήση χημικών συστατικών και με πολύ καλά αποτελέσματα και για τα ζώα και για το περιβάλλον και για τη δική μας την υγεία γιατί είναι καλύτερο να μην καταναλώνουμε χημικά συστατικά μέσω της διατροφής μας από ζωικά προϊόντα μέσω δηλαδή των ζώων και τη παραγωγή από τα ζώα. Περιορίζουμε πάρα πολύ λοιπόν την πίεση και στο περιβάλλον. Σε επίπεδο εκτροφών έχουμε γεωνομικά αποτελέσματα τα οποία είναι πραγματικά εμφανέστατα. Δηλαδή όταν μιλάμε για την, την, τροφική, την ιατρική κατάσταση των ζώων που βρίσκονται στις δικές μας εκτροφές από τη στη συμβατική κτηνοτροφία μπορούμε να είμαστε περήφανοι σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανείς μετά από ιδίως αν έχει ακούσει κανείς τα σχόλια ορισμένων. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, διότι πολλά θέματα έχουν ήδη καλυφθεί και σε, κάτι συμφωνώ, σε πολλά συμφωνώ με όσους έχουν υποθεί τώρα, αλλά εν είδη συμπεράσματος να πω ότι πρέπει να αναπτύξουμε ακόμη και όντω να προωθήσουμε την καλλιέργεια των ψυχανθών με τα σωστά κίνητρα σε επίπεδο πολιτικών, διότι ω τώρα απλώ ε, κάπω ε, μπαλώνουμε και παριστάνουμε ότι υποστηρίζουμε, αλλά δεν το κάνουμε πραγματικά ω προ την έρευνα. Οι πρωτενε ε, δεν χρειάζεται να παράγονται μόνο μέσω τη σόγια. Είδαμε τι πολιτικέ έχουν επικρατήσει ω τώρα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Υπογραμμίστηκε αυτό και σε σχέση με το τι συμβαίνει σε επίπεδο απασχόληση αλλά και κοινωνία είναι υπαρκτά τα προβλήματα αυτά. Πρέπει όμω να μελετήσουμε μια γεωργική πολιτική διαφορετική για να επιτρέψει να δημιουργηθούν θέσει εργασία και να επανέλθει οικονομική, ε, το οικονομικό πάντρεμα των τοπικών αναγκών με ε, την προστασία της υπαίθρου. Όταν χάνονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ένα τμήμα της οικονομίας που σχετίζεται με τη γεωργία επίσης χάνεται. Και αυτό αφήνει κενά. Αφήνει κενά σε επίπεδα οικονομίας και κοινωνίας. Ε, πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε και άλλο αυτό το θέμα, αλλά όπως στην περίπτωση της μυδικής και άλλων πρέ, ψυχανθών μάλλον, πρέπει να το μελετήσουμε θα πρέπει να δούμε την, ε, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μαζί με τις διατροφικές ανάγκες των ζώων και παρόλα αυτά να τονίσω ότι παραμένει ανάγκη να χρησιμοποιούμε και να εισάγουμε σόγια έστω και βιολογική, ακόμα μάλλον και βιολογική, διότι υπάρχει και ε, η ανταγωνιστική σχέση με την κατανάλωση από τους ανθρώπους. Οι καταναλωτές βιολογικών τροφίμων ε, έχουν την τάση να τρώνε πολλά προϊόντα που έχουν βασιστεί στη σόγια. Στη Γαλλία έχουμε μια παραγωγή που αρχίζει να αποκτά τον ενδιαφέρον σε επίπεδο βιολογική καλλιέργεια. Παρόλα αυτά, ακόμα υπάρχουν ε, πολλέ εισαγωγέ. Χρησιμοποιούμε παρόλα αυτά, μην το ξεχνάμε, και την ε, σόγια η οποία είναι αποφλειωμένη σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους ομιλητές για την ποιότητα των παρεμβάσεών τους και τα σχόλιά τους. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον τρίτο και τελευταίο καλεσμένο του δεύτερου τμήματο τη δημόσια ακρόαση, τον κύριο Ντέιβιτ Μακνότον, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Σόγιας Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρεία περιορισμένης Ευθύνη, Θα μας μιλήσει για τις καλύτερε λύσει για τη μείωση της εξάρτησή μα από εισαγόμενε πρωτεΐνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό σας κύριε Νότον. Έχετε πλούσια πείρα σε θέματα γεωργίας, ζωοτεχνίας. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Uh, good afternoon. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας μιλήσω για το θέμα αυτό. Η εξάρτηση από, τα από τις καλλιεργίες στην Ευρώπη είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ χρόνια τώρα. Κάνω προσπάθειες και χαίρομαι που έχει πάρει μεγαλύτερε διαστάσει τώρα. Σας πω όμως ποιος είμαι πρώτα απ' όλα. Ονομάζομαι David Μακνότν και είμαι ο ε, επικεφαλής της Soya UK ΕΠΕ. Εμπορευόμαστε δηλαδή σπόρο και ιδιαίτερα πρωτεϊνούχο σπόρο, σπόρο ειδικών τμήματων αγοράς. Λούπινα, σόγια, τριτικάλε, τριτικάλε κουκιά, μείγματα ζωοτροφών και και χρυμπάρι. Και εκπροσωπούμε επίσης ε, σπόρους για ε, λούπινα και σόγια σε άλλες χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή εκπροσωπούμε μία σειρά από ε, καλλιεργητές διαφόρων καλλιεργειών και σε αρκετές αγορές συγκεκριμένα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Εξασφαλίζουμε όλο το σπόρο λούπινο και σόγια του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά σπόρο σόγιας, φασόλι σόγιας υπάρχει. 400 εκτάρια φέτος, μηδέν πριν από δύο χρόνια. Πριν από 15 χρόνια είχαμε 1500 εκτάρια. Όμως λόγω των καταστροφικών συνεπειών της συμφωνίας Blair House. Ε, είναι πλέον αδύνατη. Η κατέστη αδύνατη η, καλή, η διατήρηση της καλλιέργειας. Εμείς μπορέσαμε να επιβιώσουμε και χωρίς υποστήριξη, αλλά μόνο μετά την αποσύνδεση. Και επίσης, όταν εμφανίστηκε σημαντική ε, εξέλιξη, αλλαγή δηλαδή στις τιμές της σόγιας. Τώρα, εξάρτηση. Ευρωπαϊκή εξάρτηση από την παραγωγή σόγιας. Για κάποιους είναι κάτι το καινούριο ίσως. Σας διαβεβαιώ όμως ότι δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Από την περίοδο που σταμάτησε να χρησιμοποιούνται, σταμάτησε να χρησιμοποιούνται για τα μερικάστικά από τον Ιανουάριο του 2001 ε, ζωοτροφές με ζωάλευρα και ηχθιάλευρα αυξήθηκε η εξάρτησή μας από τα σογιάλευρα και τότε, 15 χρόνια πριν, είχαμε εξάρτηση κατά 67% για κάθε συμπλήρωμα πρωτεΐνης που χρησιμοποιούνταν ως τροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 15 χρόνια είχαμε εξάρτηση κατά 67%. Το ίδιο επίπεδο εξάρτηση το έχουμε διατηρήσει όλη αυτή την 15 ετία. Αυτό που αλλάζει το μεταξύ όμω α και, και θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα αυτή η εξάρτηση επί 15 χρόνια. Πρέπει να αλλάξει. Επί 15 χρόνια είναι αξιών λόγου το ότι δεν ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσει το πρόβλημα. Να σας πω εγώ τι έχει αλλάξει όμως τα τελευταία 15 χρόνια. Το κόστος. Τα μετρητά. Το χρήμα. Μεταξύ 2001 και 2007 ένας τόνος σογιάλευρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κόστιζε περίπου τα 200 ευρώ. Εμείς είχαμε παραγωγή σόγια στον Ηνωμένο Βασίλειο 170 περίπου λίρες σε εγχώριο νόμισμα ο τόνος. Και είχαμε σε κάθε άριο 100 λίρες περίπου, 170 λίρες. είχαμε την απόδοση της συγκομιδής μας, 170 λίρες πώληση, αλλά το περιθώριο για το Γεωργό δεν ε, ήταν επαρκές και έτσι μας έλεγε, μα δεν με συμφέρει να καλλιεργώ τη σόγια. Είχε μικρό περιθώριο. Και αυτό βέβαια δεν ε, βοηθούσε, σε αυτό βέβαια δεν βοηθούσε το γεγονό ότι έπρεπε να φτάσουμε να κατέβουμε στα 60, σε 60 λίρε το άριο, γιατί ήταν συνδεδεμένη η σόγια με του ελαιούχου σπόρου. Τώρα, τι έχει αλλάξει από το 2008. Ότι έχει ε, εξελιχθεί φοβερά η τιμή της σόγιας. Στα τέλη του 2008, ο τόνος της σόγιας ξεπέρασε τις 300 λίρες από τις 100-150. Από το 2008 η αγορά των υδατανθράκων έχει παρουσιάσει άνοδο, κάθοδο, ξανά άνοδο και ξανά κάθοδο, ενώ η σόγια έχει μόνο σταθερή αύξηση τιμής. Σε πραγματικούς όρους η αξία της σόγιας, σε πραγματικούς όρους, η αξία της σόγιας έχει διπλασιαστεί από το 2007. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί ο Γιώργος να εξακολουθήσει να πληρώνει τέτοιο αντίτιμο για τη σόγια. Γιατί καλά να είναι καλλιεργητής. Άμα είναι κτηνοτρόφος και χρειάζεται να αγοράσει σόγια. Ναι, συγγνώμη για όλα τα νούμερα που σας έχω βάλει εδώ. Πρέπει λοιπόν να στραφούμε στο μέλλον. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Νομίζω σε πολύ απλούς όρους μπορώ να σας τα πω όλα με βάση αυτή τη διαφάνεια. Η απάντηση είναι όχι, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Το κόστος της σόγιας θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η κατανάλωση σόγιας όλο τον κόσμο θα ξεκολουθήσει να ενισχύεται, ίσως με βραδύτερους ρυθμούς. Η παραγωγή της σόγιας παγκοσμίω ήδη έχει σημειώσει ε, δραματική αύξηση, σημαντική αύξηση. Η γεω φυτικές ε, βελτιώσεις και γενετικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, πραγματοποιήθηκαν. Στην Αμερική, Αμερικανική Ήπειρο έχουμε ε, τεράστια ενίσχυση της, αύξη, ενίσχυση της παραγωγής και νέες ποικιλίε ε, χάρη στα γενετικά τροποποιημένα. Τεράστιο αριθμό, δηλαδή δεν αναμένεται να υπάρχει αντίστοιχο άλμα στην παραγωγή και τη συγκομιδή η ε, εμφάνιση νέων ποικιλίων σόγια στην επόμενη 15 αιτία, αλλά οπωσδήποτε θα αυξηθεί η κατανάλωση σόγια στην επόμενη 15 αιτία. Αυτό ναι θα το δούμε γιατί θα συνεχίσει η κινέζικη αγορά να αγοράζει όλο και περισσότερη σόγια. 75 εκατομμύρια μέχρι 80 εκατομμύρια τόνους καταναλώνει αυτή τη στιγμή η κινέζικη αγορά. Δεν είναι καθόλου απίθανο στην επόμενη 15 ετία να έχουν, ε, να έχουν αρχίσει να συσσωρεύουν εκατοντάδες εκατοντάδες τους τόνους της σόγιας στην αγορά από την αγορά οι Κινέζοι. Αν συμβεί αυτό, το κόστος για τον κτηνοτρόφο από την εξασφάλιση ε, πρωτεϊνούχου ζωοτροφής για τα ζώα του θα ε, καταστεί δυσβάσταχτο. Και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι ομιλητές σήμερα αποδέχθηκαν ότι είναι παράλογο αυτό το επίπεδο εξάρτησης και ο Μαντίας μας είπε ότι έχουμε να κάνουμε ένα προϊόν εισαγόμενο και πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση. 185 λίρες το εκτάριο κοστίζει στον γαλακτοπαραγωγό της Αγγλίας η αγορά των ζωοτροφών. Δεύτερο μόνο στη σειρά είναι το κόστος του εργατικού δυναμικού. 90 λίρες το εκτάριο. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόστος και κατά το διπλάσιο είναι αυτό της αγοράς των ζωοτροφών. Και είναι η επιβάρυνση αυτή μόνη για την αγορά, για την εξασφάλιση της πρωτεΐνης και όχι για προσθεμένη αξία κάτι. Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, και σας το λέω να μην έχετε καμία ψευδέστηση, ε, ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει κέρδος, δεν παράγει κέρδος ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος της Ευρώπης σήμερα. Γιατί, Γιατί έχει κόστος και τεράστιο, με μεγάλη διαφορά δηλαδή, κόστος μεγάλο ε, στην εξασφάλιση της πρωτεΐνης. Ε, ποιος ρώτησε νωρίτερα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε μια πολυτομεακή προσέγγιση. Πρώτον, συμφωνώ ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή της σόγιας στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να γίνει με την ε, αναγκαστική αδειοδότηση των μεταλλαγμένων Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχει δυναμικό συγκομιδής, ενίσχυση συγκομιδής από το μεταλλαγμένο στο μη μεταλλαγμένο στο 5% ανεξαρτήτως των εγγενών χαρακτηριστικών του μεταλλαγμένου, τα οποία γεννή χαρακτηριστικά με τις τέσσερις ποικιλίε που έχουμε, μόνο ε, ανθεκτικότητα σε ε, μπορούν να προσφέρουν. Δεν χρειαζόμαστε τα μεταλλαγμένα. Ναι, μπορεί να έχουν κάπως μεγαλύτερη απόδοση ε, τα μεταλλαγμένα. Αλλά δεν τα χρειαζόμαστε. Κάποιοι λένε ότι για να λύσουμε τα προβλήματα ω προ την εξασφάλιση πρωτεΐνης στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μεταλλαγμένα. Όχι, είναι ανοησία αυτό. Πραγματικά δεν ισχύει. Πρέπει να μέγιστοποιήσουμε την παραγωγή τη όγια η αξία του ή να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή αρακά και φασολιού και ιδιαίτερα θέλω να δώσω τη σημασία της πρωτεΐνης του αρακά και του φασολιού. Είναι χαμηλή τεχνολογία η παραγωγή του αρακά, δεν ξέρω γιατί δεν παράγουμε περισσότερο. Και όπως είπε και ο φίλος από εδώ, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις φυσιφιστάμενες πηγές ε, πρωτεϊνών, τριφύλλη, μυδική, ό,τι άλλο υπάρχει πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Πρώτα λοιπόν τις βασικές, τα βασικά πρωτεϊνούχα ε, για να έχουμε μία βάση και μετά με φασόλια και αρακά μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο. Ξέρω ότι έχω περάσει το χρόνο μου, αλλά μπορούσα να σας πω πόσο καταπληκτική καλλιέργεια είναι τα λούπινα. Εγώ χρόνια τώρα τα καλλιεργώ. Είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε περισσότερο. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το, χώρο το χρόνο μου. Συμφωνία Blair House. Βεβαίω πρέπει να συζητήσουμε το θέμα τη συμπερίληψη τη σόγιας ε, στα καθεστώ των ελαιοχών. Θα χρειαστεί ασφαλώ επανα διαπραγμάτευση των συμφωνιών της ΓΑΤ, ε, αλλά νομίζω ότι για να ενισχύσουμε το πρασίνισμα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνουμε σε αυτό και να προχωρήσουμε και βεβαίως χρειάζεται ένα σύστημα, όπως είπε και ο Δ. Καζαούσκη, με ε, κίνητρα ανταπόδοση, αναγνώριση της ενεργειακής αξίας που μας εξασφαλίζουν ε, τα ψυχανθή χάρη στην συγκράτηση των αζωτούχων ενώσεων. το ισοζύγιο των ψυχανθών και οσπρίων ως προς την ε, ε, συγκράτηση των αερίων θερμοκηπίου είναι πολύ καλύτερο από αυτό των λεγόμενων ενεργειακών καλλιεργείων. Γιατί λοιπόν να μην δώσουμε επιδότηση σε, αυτά, σε αυτές τις καλλιεργίες. Από το 1992 δεν έχουμε δώσει τέτοια ενίσχυση στα ε, όσπρια από τη στιγμή που σταμάτησε η διαδικασία ε, η επιδότηση επεξεργασίας ή καταργασίας ε, αρακά και φασολιών δεν υπάρχει καμία στήριξη για αυτά ε, τι καλλιέργειες. Προφανώ προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα που σωστούμε Και έτσι λοιπόν κλείνοντα, σα ευχαριστώ πολύ. Να και ένα ωραίο λιβάδι με λούπινα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου σήμερα, γι' αυτό και είμαστε πιο χαλαροί στην χορήγηση χρόνου ομιλίας. Δεν έχουμε τόσο πιστικό πρόγραμμα στην ημερήσια διάταξη όπως συνήθως. Γι' αυτό και δεν σας διακόπτω, ούτε είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση του χρόνου. Και τώρα περνάμε στη συζήτηση μετά το δεύτερο γύρο, ε, το δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόσης. Πρώτη ζήτησε το λόγο η κυρία Αγγιλέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω συγκεκριμένη ερώτηση προς όποιον θέλει να απαντήσει. Είμαι Ισπανίδα και όντως ε, η στήριξη της ΚΑΠΑ στα ψυχαθή ήταν ελάχιστη. Εξού και εξαφάνιση αυτών των καλλιεργειών. Στην Ισπανία δεν είχαμε καμία τέτοια ενίσχυση για τα ψυχαθή, δυστυχώ. Πιστεύετε λοιπόν ότι στη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μπορούμε να ε, περιλάβουμε στις ενισχύσεις του πρασινίσματος σε κάποια, ε, να περιλάβουμε κάποιες ενισχύσεις όχι για τα τα βιολογικά, αλλά στα πλαίσια του greening μια ενίσχυση για τα ψυχανθή, γιατί δεν είναι όλα βιολογικά ή οικολογικά τα προϊόντα. Είναι ενδιαφέρουσε και οι βιολογικέ παραγωγέ, αλλά θα μπορούσαμε μέσω του, του κεφαλαίου για το πρασίνισμα να στηρίξουμε τι καλλιέργειε ψυχανθών. Επίση, τι αντίκτυπο έχουν οι συμφωνίε με τρίτε χώρε στην παραγωγή σόγιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί σίγουρα και αυτές οι εμπορικές συμφωνίες συνέβαλαν στην απόλυτη εξάρτησή μας από την εισαγόμενη σόγια. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή σόγιας, κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Σέρτος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για τον ε, Ματσία Σκιώνα έχω μια ερώτηση. Ποια είναι η ενδεχομένη θετική εμπειρία που έχετε από τις ενώσεις σας ενός παραγωγών και πού βλέπετε κάποιες ελλείψεις ενδεχομένω. Τι λείπει, τι θα θέλατε να δείτε να συμβαίνει περισσότερο και τι γνώμη έχετε για την ε, ε, παραγωγή ζωοτροφών χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σοραπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα της παραγωγής ε, πρωτεϊνούχων φυτών ε, είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο και θα παραμείνει επίκαιρο και στο μέλλον. Γιατί όσο περισσότερο παράγουμε και όσο λιγότερο εισάγουμε στην Ευρώπη, τόσο καλύτερη θα είναι η κατάστασή μας. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα τώρα, για να ενταθεί η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών. Θα μπορούσαμε ως κίνητρο να στοχεύσουμε προς τους πελάτες, δηλαδή τους καταναλωτές, να δώσουμε κίνητρα στους καταναλωτές για να αγοράζουν ε, φυτική πρωτεΐνη κοινοτικής παραγωγής, ε, ευρωπαϊκής παραγωγής. Στη Λιθουανία είχα μια σειρά συναντήσεων με παραγωγούς και ανακάλυψα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι δικοί μας καλλιεργητές, η δική μας παραγωγή ισχυρίζονται ότι έχουν δυσκολίες ε, με την ε, ετικετοθεσία των προϊόντων ως απαλλαγμένων από μεταλλαγμένους οργανισμούς, γιατί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν δικαιούνται να δώσουν αυτό το σήμα. Θα πρέπει να στείλουν επίσημη επιστολή και έχουν πρόβλημα γενικώ με τη σήμανση των προϊόντων τους ως ε, απαλλαγμένων από μεταλλαγμένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια κριτήρια και κάποιου ε, όρους και απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, η, η γάλακτοπαραγωγή που δεν χρησιμοποιούν ζωοτροφές με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς για τα ζώα τους, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, GMO-free. Ευχαριστώ. Κύριος Φλάνεγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν να πω ότι είναι από τις καλύτερες αυτή που άκουσα του κύριου Μακνάδου. Πολλά έμαθα, είναι πολύ ενδιαφέροντα και βλέπω ότι τη ε, δουλειά σα την κάνετε με πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάθος να το συνεχίσετε λοιπόν. Δύο χρόνια που είμαι εδώ, πρώτη φορά βλέπω τέτοια παρουσίαση. Ε, τώρα, το πώς μπορούμε να περάσουμε από τη σόγια σε άλλου ε, πρωτεϊνούχου καρπού, ότι δηλαδή το ένα πρωτεϊνούχο είναι ισοδύναμο με ένα άλλο πρωτεϊνούχο, είναι με το πετρέλαιο, είναι ισοδύναμο με το νερό, είναι και τα δύο υγρά και άρα μπορούμε να, να τα χρησιμοποιήσουμε υπελακτικά. Ε, δεν νομίζω ότι έχουν όλα αμινοξέα στην ίδια γκάμα και πολλά από αυτά που λέγονται σήμερα φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ε, αν θέλω να κλειτώσω από τη σόγια δεν ε, χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο παρά να ε, βρω μια άλλη πρωτεϊνούχα καλλιέργεια. Αλλά δεν, δεν είναι δεδομένο ότι έχει και η άλλη καλλιέργεια αυτή της, της, τα ίδια συστατικά, τις ίδιες ουσίες να προσφέρει. Φέρει το λούπινο το οποίο αναφέρατε και φαίνεται ότι θα γίνουμε φανατικοί υποστηρικτές του. Έχει πράγματι, μπορεί να είναι εντελώς ισοδύναμο με τη σόγια. Ευχαριστώ κυρία Πέτυρ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είχαμε ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, γι' αυτό έφτασα πιο αργά. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου και το θαυμασμό μου για την παρουσίαση του κυρίου Μακνότον, γιατί πραγματικά συνόψισε πολύ εύστοχα το μεγάλο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών. Ε, είμαι από την Κροατία είμαστε χώρα χωρίς ε, μεταλλαγμένους οργανισμούς, δεν επιτρέπουμε τη χρήση γενετικών τροποποιημένων οργανισμών και μάλιστα ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία σόγια του Δούναβη για να ε, παραγάγουμε αρκετή σόγια ώστε να γίνουμε αυτάρκη σε σόγια, πάλι στα μη μεταλλαγμένη σόγια, αντί να χρησιμοποιούμε εισαγόμενη σόγια που δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της και αν είναι μεταλλαγμένη ή όχι. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παράγουμε επαρκή σόγια αλλά και ε, άλλες πρωτεΐνες από ψυχαθή, όσπρια, ε, μπιζέλια και ούτω καθεξής. Συμφωνείτε ότι είμαστε αρκετά ικανοί για να κάνουμε κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε αυτή η χρονιά ήταν η χρονιά των οσπρίων. Ε, γιατί είναι σημαντικά τα όσπρια όχι μόνο για την ανθρώπινη διατροφή αλλά και για την διατροφή των ζώων, για τις ζωοτροφές. Μπορούμε λοιπόν κατά τη γνώμη μου να καταλήξουμε σε αυτάρκεια ε, στην παραγωγή πρωτεΐνης και για τα ανθρώπινα τρόφιμα και για τις ζωοτροφές και μάλιστα χωρίς μεταλλαγμένους οργανισμούς για την παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών. Συμφωνείτε μαζί μου, ευχαριστώ. Κύριος Χόισλινγκ. <coughs> Ναι, πράγμα θέλω να το μιλήσω την κλιματική διάσταση κατά την καλλιέργεια ε, ψυχανθών. Νομίζω ότι αν κοιτάξουμε αυτή την ε, πτυχή, αν δούμε δηλαδή τι κερδίζουμε από την εξοικονόμηση διοξιδίου του άνθρακα, ε, επίσης ε, αζωτούχων ενώσεων, ε, από κατανάλωση των υδρογονανθράκων, δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια τιμολόγηση το ΣΥΠΗΝ με κλιματικά πιστοποιητικά για τα ψυχανθή. Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε να προσφέρει η γεωργία στην υπόθεση της κλιματικής αλλαγής. Και κρίμα, κατεβάσατε την ε, διαφάνεια για τα λούπινα χωρίς να μας δώσετε λεπτομέρειες. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ακριβώς ποια είναι τα πλεονέκτηματά τους σε σχέση με την καλλιέργεια της σόγιας, γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για πολλές περιοχές. Είπατε ότι δόθηκε ιδιαίτερη όθηση με την αποδέσμευση των πληρωμών. Νομίζετε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξουν πάλι συνδεδεμένες πληρωμές για να δώσουμε μια νέα όθηση. Και καταλήγοντα, θα ήθελα να πω ότι ναι, συμφωνούμε. Είναι πολλά και λογικά τα μέτρα που θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε, η λύση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά ερωτώ γιατί δεν γίνεται τίποτα. Ποια είναι αυτή η ομάδα των λόμπι που εμποδίζει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αφού χρόνια τώρα Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μποϊκοτάρουν εσκεμένα και δεν δέχονται παραδείγματι να μπουν στην αγορά συγκεκριμένες πρωτεϊνούχες παραγωγές συγκομιδές όπως ε, τα λούπινα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη. Ε, euh, euh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, ομιλητές. Πρόεδρε, δεν σας κάνω εύκολα φιλοφρονήσεις, αλλά είναι σημαντικό που προβλέψατε αυτή τη συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας από την επικαιρότητα και ευχαριστώ και όλους τους ε, ομιλητές, κυρίως την κυρία Λεπελετιέ, η οποία καλό είναι να ακούγεται, μαζί με άλλους Γάλλους που εκπροσωπούν κοινοτρόφους και γεωργούς. Όπως είπε και ο κυρίος ε, Λουαζό, για, από την πλευρά των γεωργών, καλλιεργητών θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση της Ευρώπης και της Γαλλίας στη σόγια, που εισάγουμε σε μεγάλες ποσότητες. Θα πρέπει να ανακτήσουμε την αυτάρκειά μας ως προς τη σχετική παραγωγή. Σήμερα η παραγωγή της σόγιας είναι 1% η ευρωπαϊκή παραγωγή σόγιας είναι 1% των αναγκών των, της ευρωπαϊκής κοινοτροφίας. Και για άλλη μια φορά οι συμφωνές, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, εμπορίου, κυρίως με τις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά. Αυτές επικρατούν και ε, κάνουν ε, ένα εμπορικό προϊόν ε, και τα δημητριακά ιδίως για τη σόγια μας έχουν στο χέρι οι χρηματαγορές. Για τις χώρες που κυριαρχούν εδώ, ξέρουμε ποιες είναι στις αγορές, αλλά θα πρέπει λίγο να πάρουμε αποστάσει από αυτέ τι ε, συμφωνίε του το και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει τη δική τη της σόγια χωρί να πέφτει στα γρανάζια των μεγάλων βιομηχανικών ε, εταιριών που ε, απειλεί και την αυτοκυριαρχία τη Ευρώπη και την δική μα βιομηχανική παραγωγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο μιλητή. Εξαντλήθη ο κατάλογος. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας, στους καλεσμένους μας, με τη σειρά που μίλησαν και προηγουμένως. Ο κύριος Κρέων είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής ε, για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και τα σχόλιά τους. Ανακεφαλώνοντας τη συζήτηση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ μπορώ να σας παραθέσω τη δική μου εμπειρία και τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της σόγιας. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που θα είναι προσανατολισμένη προς την αγορά. Και μάλιστα εμείς έχουμε επιστοποίηση στην οργάνωση. Το Danube Soja είναι το σήμα που δίνουμε, σόγια του Δούναβη και μπορούμε να το αναφέρουμε σε προϊόντα γαλακτοκομικά που περιέχουν ζωοτροφές ή σόγια που χρησιμοποιήθηκε από εμά που είναι μη μεταλλαγμένη, είναι βέβαια λίγο πιο ακριβή από τη βραζιλιάνικη σόγια, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε μια κατεύθυνση, ένα προσανατολισμό προ την αγορά. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη σόγια, ισχύει και για τα άλλα ψυχανθή. Ε, σίγουρα η ντόπια παραγωγή είναι πιο ελκυστική και αν ε, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι θέλουν να, να έχουν τοπικές ζωοτροφές, χώρες ζωοτροφές, θα πρέπει να τις παράγουν τοπικά και νομίζω ότι έτσι δημιουργείται ένας πολύ θετικός, σενάριο κύκλος εγκύτητας, ώστε θα έχουμε πρώτες ύλε για ζωτροφές στην χώρα και με τόπιες ζωτροφές θα εκτρέφονται τα ζώα, κάτι που δημιουργεί μια πολύ θετική εικόνα. Και αν θέλουμε ε, ψυχανθεί, δεν αρκεί να τα καλλιεργούμε μόνο, αλλά θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε στα προϊόντα, και να τα διαθέτουμε και στην αγορά. Εμείς είμαστε μία ένωση, μία οργάνωση που προσανατολίζεται προς την αγορά μας. Ενδιαφέρει και η εμπορευματοποίηση. Και δεν έχουμε καμία στήριξη δημόσια. Είμαστε ιδιωτική ένωση. Επίσης θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν άλλο κύκλο για τα ψυχανθή, να ξεπεράσουμε αυτό το φαύλο κύκλο που έχει δημιουργηθεί, να δώσουμε ενάσματα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε οι πρωτεϊνούχε και ελαιούχε παραγωγέ να γίνουν πιο προσοδοφόρες για τον Γεωργό. Κάτι που δεν ισχύει. Ε, ο κόσμος έχει αρχίσει να ζητά και ευρωπαϊκή σόγια και αρχίζουν οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, για καλύτερου σπόρους σόγια και ίσω μετά από μια δεκαετία θα έχουμε περισσότερη ευρωπαϊκή σόγια και θα είναι προσοδοφόρα ε, οικονομικά. Αλλά για άλλε καλλιέργειε, τα λούπινα, τα πίσα, τα μπιζέλια, ο κόσμο δεν έχει την αίσθηση ότι θα, ε, θα αναπτυχθούν αυτέ οι παραγωγέ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, τροφοδοτήσει αυτήν την εντύπωση ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιου είδου πρωτεϊνούχε παραγωγέ. Σίγουρα πρέπει να έχουμε μια πενταετία ε, τώρα η δαμόκλος πάθη επικρεμάται πάνω μας. Ε, δημιουργείται μια ανασφάλεια όταν δεν έχουμε ένα προβλέψιμο ορίζοντα και δύσκολα θα γίνουν και επενδύσεις χωρίς τέτοια προβλεψιμότητα. Καλές είναι και οι δημόσιες επενδύσεις, αλλά δυστυχώς περιορίζονται μόνο στη βασική θεμελιώδη έρευνα. Εμείς χρειαζόμαστε και πιο προηγμένη έρευνα και αυτό θα προέλθει από ιδιωτικέ επενδύσεις. Θα πρέπει να έχουμε συντονισμένη προσπάθεια και σε βάθος χρόνου για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θέλουμε μια ασφάλεια του σχεδιασμού. Αυτό είναι σημαντικό. Εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για το μέλλον. Και έτσι δημιουργείται ένα ενάρετο κύκλο επενδύσεων στι καλλιέργειε και οι καλλιέργειε γίνονται και πιο οικονομικά βιώσιμε και προσοδοφόρε. Επίση, να δώσουμε κίνητρα για την ζήτηση με σήμανση των προϊόντων και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα ασφάλεια του σχεδιασμού για τι εταιρείε. Και δηλαδή να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα ψυχανθή όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα και συνεχώς. Ευχαριστώ. Κύριε Πελετιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω στο θέμα της σόγιας, διότι δίνεται εντύπωση ότι χωρίς τη σόγια δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε και να καταργήσουμε, δεν χρειαζόμαστε. Χρειάζεται μια σχετική ισορροπία, όμως εδώ και κάποια χρόνια Διαρκώς ε, μιλάμε για τη σόγια, λες και είναι το μόνο που, προϊόν που μπορούμε να έχουμε. Ήδη στη συμβατική κοινοτροφία είναι πολύ σημαντικό προϊόν και στην αναλογία φτάνουμε το 40, 60 ή 80% σόγιας στην περιεκτικότητα. Είναι πραγματικά ε, φοβερό αν δουλεύει κανείς ως προς την υγεία ή την ευζοία των ζώων έχει πρωτεΐνες σίγουρα, αλλά τα αμινοξέα στη διατροφή των ζώων μπορούμε να τα πάρουμε και από αλλού. Όπως έλεγα στις φρόμουλες που χρησιμοποιούμε, δεν έχουμε πάρα πολλά αμινοξέα βιολογικά, δεν είναι πολύ διαθέσιμα, αλλά την καλή διατροφή των ζώων την πετυχαίνουμε με άλλα τεχνικά μέσα και τα ανάλογα αποτελέσματα, τα μονοξέα. Είναι σημαντικά για του χείρου και τα πολυερικά και τα βρίσκουμε από τα ψυχανθή κάποιε φορέ. Η ισορροπία είναι πραγματικά επίση <clears throat> πολύ καλή. Οι μονοκαλλιέργειες νομίζω ακόμη έχουν δείξει τι μπορούν να προσφέρουν. Δεν φέρνουν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Και όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα, για καλλιέργειε που μπορεί να είναι ποικίλε σε επίπεδο τη ίδια εκμετάλλευση, καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο χημικά συνθετικά προϊόντα από την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε, να απαλλαγούμε από αυτά. Μπορούμε να τα μειώσουμε δραστικότατα. Αυτή τη στιγμή υπάρξει απαραίτητη ποικιλία. όταν κάποιο καλλιεργεί λόγω χάρη μανιτάρια και θέλει ανάλογες ε, ε, σοδιές, ποσότητες σοδιάς και χρησιμοποιεί νικητοκτόνα, μπορεί να αλλάξει αυτό τον κύκλο με την αναλλαγή της καλλιέργειας και να έχει επίσης γεωργικούς κύκλους ε, σοδιάς πολύ ικανοποιητικού. Πρέπει λίγο την δική μας την αντίληψη να βλέπουμε την γεωργία και την κτηνοτροφία εδώ και κάποια χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο να την μεταβάλουμε. Ε, βλέπουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το που φτάσαμε. Μιλήσατε προηγουμένω για τα προβλήματα τη αγορά εργασία. Όντω, όταν μιλάμε για μεσαίε εκμεταλλεύσει και δουλεύουν αυτέ με κάποιε συγκεκριμένε ε, εκτροφέ, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε και τους αριθμούς που θέλουμε. Γιατί αν σκεφτούμε και τι κοινωνικέ τις από τη σκοπιά τη κοινωνία, κάποιε αλλαγέ πρέπει να γίνουν. Πρέπει να εργαστούμε επίση στο τοπικό επίπεδο. Όταν λέμε ότι δεν έχουμε αρκετό κέρδο και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξάγουμε, α κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να ξανακατακτήσουμε την εσωτερική αγορά. Εκεί μπορούμε να βρούμε ίσω ήδη μια ισορροπία. Είμαι πεπισμένη ότι, όπως έλεγε προηγουμένως ε, και ο συνάδελφος, δεν μπορούμε να πετούμε βιολογικές καλλιέργειες παντού, όμως πληροφορίες για αυτό το είδους τη γεωργία και αυτό το είδους τη διατροφή που έχουν δώσει αποτελέσματα, να τις συγκεντρώσουμε και να δούμε πώς με καλύτερο τρόπο μπορούμε να τροποποιήσουμε και να αλλάξουμε την κατεύθυνση της γεωργίας και της τεχνοτροφίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Νότον. Μακνότον. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει 25 με 30 τόνους σόγιας και σόγια ολευρού από την παγκόσμια αγορά κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Το θέμα είναι ότι αντιστοιχεί στο 65 της πρόσθετης σόγιας. Και αν σταματήσουν αυτά τα πλοία να φτάνουν εδώ, από την Αττινική Αμερική, τι θα γίνουν και τα χειροστάσια και τα ε, εργοστάσια πουλερικών, οι μονάδες πουλερικών κτλ. Σε τρεις μήνες να σταματήσουν. Από τώρα να σταματήσουν σήμερα. Σε τρει μήνε θα είμαστε σε πολύ δεινή κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί εξαρτώμεθα λοιπόν τόσο πολύ και γιατί, γιατί δεχθήκαμε να εξαρτηθούμε τόσο πολύ τα τελευταία 15-20 χρόνια. επεσήμανε ο κύριος Φλάνναγκαν πολύ σωστά ότι η απάντηση έχει να κάνει με το προφίλ αμινοξέων είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των θιούχων αμινοξέων της σόγιας που φέρνουν περισσότερη ενέργεια στα σύγχρονα ζώα, χείρο, κοτόπουλο και το καθεξής λαϊκίνη και μεθαϊονίνη χρειάζονται για να παράγουν κρέας. Λαϊκίνη πάνω απ' όλα. Για την παραγωγή του γάλακτος χρειάζονται μεθαϊονίνη. Μεθιανίνη. Πρόκειται για θείου με ιδιαίτερη υψηλή παρουσία στη σόγια. Και γι' αυτό για να έχουμε υψηλού επίπεδο, υψηλού επίπεδο παραγωγή κτηνοτροφική, κοτόπουλα με πολύ κρέας κτλ. δεν μπορούν να τους προσφέρονται πρωτεΐνες, χαμηλ, πρωτεΐνες χαμηλής απόδοσης γιατί δεν θα έχουν την απόδοση που απαιτεί η σύγχρονη εκτροφική μέθοδος. Το σύστημα λοιπόν δεν θα είναι εύκολο να το ανατρέψουμε γιατί είναι αλληλένδετη η γενετική των ζώων με το είδος καυσίμου που θα χρειαστούν. Δεν μπορεί να βάλει κανείς ε, σε μηχανή ενός ε, αεροπλάνου ε, αεριοθούμενου δίζελ. Το ίδιο είναι αυτό που σας λέω τώρα. Τα σύγχρονα αυτά ζώα είναι σαν μεταβολικά αεριοθούμενα. Χρειάζονται συγκεκριμένο καύσιμο. Αυτό το καύσιμο το προσφέρει η σόγια η μόνη άλλη καλλιέργεια. Και ευχαριστώ που μου, το, μου δώσατε και την ατάκα κύριε ε, Χόισλινγκ. Είναι ακριβώς το λούπινο με υψηλό κατά 40 περίπου της υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και άρα είναι συγκρίσιμη. Το σογέλαιο 44-47% ανάλογα τι αγοράζει κανείς. Το λούπινο έχει 40. Ο αρακάς του φασόλι στα 25 περίπου. 100. Γι' αυτό το λούπινο μπορεί να ανταγωνιστεί. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια επίπεδα ποιότητας που πρέπει να διατηρηθούν και για την ε, ζωική παραγωγή. Αυτό εξηγεί άλλωστε και την, αυτή η, η απέτηση σε υψηλή ποιότητα σε πρωτεΐνη ε, εξηγεί γιατί εξαρτώμεθα τόσο πολύ από την εισαγωγή σόγιας. Δεν μπορούμε ξαφνικά να σταματήσουμε τη σόγια και αρχίσουμε να τους ε, να τους δίνουμε φασόλια και αρακά. Δεν, δεν, δεν θα αρκούσε κάτι τέτοιο. Μόνο με το λούπινο μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη σόγια. Θα έπρεπε να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλη και εκτεταμένη παραγωγή της του λούπινου όπως της σόγιας. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό, γιατί τα πραγματικά αγρονομικά προβλήματα τα σχετικά με το λούπινο τα ξεπράσαμε μόνο μέσα στη τελευταία δεκαετία. Και για να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό, της ε, αποδέσμευσης ή επαναδέσμευσης, επανασύνδεσης. Θα σας εξηγήσω το εξής, ότι ένα από τα προβλήματα της Σόγια στην Ευρώπη ήταν το εξής, ήταν, είχε την ατυχία το 1992 η σόγια να μπει μέσα από τη συμφωνία Blair House στην κατηγορία μαζί με τους ελαιούχους πόρους και ο Ματής θα σας εξηγήσει πόσο τεράστια προβλήματα προέκυψαν από αυτό. Τεράστια προβλήματα να σας το εξηγήσω και αλλιώ 93-94. Εγώ μπορούσα να πω σε έναν ε, Γιώργο, δεν πας να φυτέψεις λίγη σόγια. Μα μου λέει 120 λίρες το εκτάριο, επιδότηση, ελαιούχη, 180 ορακάς και τα φασόλια που έχουν μπει στο καθεστώς των πρωτεϊνούχων. Ενώ ατυχώς πώς είχε δεσμευτεί μέσα στην ομάδα των ελαιούχων η Σόγια. Και αυτό εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούσε να προχωρήσει αυτή η καλλιέργεια της σόγιας στην Ευρώπη μέχρι ότου ανέβηκε πολύ τιμή της. Τα τελευταία 5-6-7 χρόνια το πολύ. Έχει οικονομική αξία, οικονομικό συμφέρον για την καλλιέργεια στην Ευρώπη η σόγια. Μέχρι τότε δεν άξιζε. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε, πώς ορθώνουμε αυτό το, αυτή την παράλογη εξάρτηση. Είμαστε τρεις μήνες μπροστά από μια καταστροφή. Επίσης, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, θα, οι Κινέζοι θα αρχίσουν να τραβάνε από την αγορά μέσα στην επόμενη πενταετία και 100 τόνους ακόμη. Πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Δεν έχουμε φτάσει στον το, δεν, δεν έχουμε φτάσει στα όρια της κατάστασης ανεβαίνουμε ακόμα. Πρέπει τώρα να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Και πρέπει να μειώσουμε τις εξαρτήσεις, την εξάρτησή μας. Έχω εξετάσει κάθε δυνατή λύση. Η πιο νομίζω πρόσφορη και αφήνω τα γενετικά τροποποιημένα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εξάρτηση 30 εκατομμύρια τόνοι. Τι χρειάζεται, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική για τι πρωτεΐνες, για τους πρωτεΐνους και τις καλλιέργειες. Εδώ στην Ευρώπη μία η οποία θα ενσωματώνει και τα λούπινα με τη σόγια και τα ψυχανθή και τους αρακάδε φασόλια μέσα σε μια ολοκληρωμένη πολιτική αυτές τις τρεις κατηγορίε, Γιατί αν μπορέσουμε αυτέ τι τρει ε, καλλιέργειε να τι. Ε, όργανο να τις προωθήσουμε κατά τρόπο ενοποιημένο, τότε μπορούμε να δώσουμε απάντηση στην εξάρτηση από τη σόγια, στις εισαγωγές σόγιας. Και για να απαντήσω στην ερώτηση σας πώς προχωρούμε σε ανεξαρτητοποίηση ως προς τις εισαγωγές σόγιας, η απάντηση είναι αυτή. Και τα ψυχανθή. Και ο αρακάς φασόλιο. Και τα λούπιτα μαζί με την εγχώρια σόγια πρέπει να μέσα από μια ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη πολιτική να αναγνωριστεί σε ποιο βαθμό συμβάλλουν και σε τι συμβάλλουν. Αυτά όλα που αναφέρθηκαν όταν είναι σωστά. Ένα μοντέλο ε, επί παραδείγματι αξιολόγηση των συνεπειών σε εκπομπέ άνθρακα είναι πάρα πολύ σωστή πρόταση. Και είναι ίσως η κατάλληλη πρόταση, αν σκεφτείτε δύο λίτρα φυσικού αερίου χρειάζονται για τρία κιλά ε, νητρικού αμμονίου, ενώ χρειάζεται καύσιμο υγρό, ορυκτό καύσιμο, σε τεράστιες ποσότητες. Η σόγια χρειάζεται 200 κιλά στο εκτάριο, 90 λίτρα δίζελ ουσιαστικά. Ο υπολογισμός ενεργειακός είναι πολύ καλύτερος από οποιαδήποτε ενεργειακή καλλιέργεια μπορούμε να ενισχύουμε με χρήμα του Ευρωπαίου ε, φορολογουμένου. Λάθος καλλιέργειες ε, υποστηρίζουμε αν θέλουμε και να σώσουμε τη διατροφική αλυσίδα μας και να σώσουμε τον πλανήτη ε, πρέπει να στραφούμε προς αυτές τις τρεις ομάδες καλλιεργειών. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι με την προσέγγιση αυτή των φυτικών πρωτεϊνών ε, όλοι τα τους επενούμε, έχουμε ενθουσιαστεί στη θεωρία, αλλά στην πράξη προτιμούμε τη γεωργία μεγάλης κλίμακος και οι πολιτικές αποφάσεις ε, ε, που λαμβάνονται δεν στηρίζουν οικονομικά αυτές τις καλλιέργειες. Παρόλο που ως προς τη θεωρία συμφωνούμε όλοι ότι είναι το ζητούμενο. Θα το δούμε πάντως και στη συνέχεια αυτό το θέμα στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης της ΚΑΠ και της μελλοντικής μεταρρύθμισης. Σας ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε όλους τους καλεσμένους μας για τις παρουσιάσεις που έκαναν. Πολύ χρήσιμες. Και σημαντικές και οι προτάσεις τους και οι συστάσεις τους. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ε, συναδέλφους που έλαβαν μέρος στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελεί σημαντικό τμήμα της ε, αηφόρου γεωργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του ευρωπαϊκού διατροφικού μοντέλου. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία, την αηφορία και την βιοπικιλότητα και το μεγάλο, την αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού που έχουν αυτές οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισορροπημένη προσέγγιση, όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική, όπως είπατε κι εσείς, ώστε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη αυτάρκεια χάρη στην οικονομική και πολιτική στήριξη αυτών των πρωτενούχων καλλιεργειών. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και πάλι τους εμπειρογνώμονές μας Έχουμε ένα ακόμη σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αν έχετε χρόνο μπορείτε να παραμείνετε για να το συζητήσουμε. Πάντως είμαστε ευγνώμονες στους εμπειρογνώμονες για τη συμμετοχή τους. Περνάμε στο σημείο 10, βιολογική παραγωγή και σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Όπως ξέρετε, έλαβε χώρα ένας ακόμη τριμμένης διάλογος, ο έβδομος επί Ολλανδικής Προεδρίας, Ο τελευταίος τριμέρης διάλογος έγινε στις 16 Ιουνίου. Δυστυχώς ε, δεν ε, διεκπαιρεώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα μεταβιβαστεί στη Σλοβακική Προεδρία. Και ευχαριστώ θερμά την, ε, τον εκπρόσωπο της Σλοβακικής Προεδρίας που είναι πάνω στην αίθουσα και θα παρακολουθήσει τη συζήτηση. Δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Χόισλινγκ, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ευχαριστώ και πάλι τους καλεσμένους μας ε, και τους χαιρετώ. Κύριε Χόισλινγκ, σας ακούμε. Ναι, πρόεδρε, το είπατε κι εσείς. Ολοκληρώσαμε την ένατη συνεδρία στο Μερός Διαλόγου την προηγούμενη εβδομάδα. Οφείλω να ευχαριστώ θερμά την Ολλανδική Προεδρία για τις σημαντικές πρόοδους που έχουμε εξασφαλίσει σε ένα θέμα καθόλου. Απλό, βιολογικές καλλιέργειες, βιολογική παραγωγή. Θα μου πείτε γιατί δεν κλείσαμε τα θέματα. Ε, τραβάει πολύ υπόθεση, το ξέρω αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ με την Ολλανδική Προεδρία. Εγώ έτσι τα αξιολογώ. Εγώ τα πράγματα άλλο μπορεί να μου πει, Α, είναι άδειο το ποτήρι. Εγώ θα πω ότι είναι μισό γεμάτο. Ευχαριστώ την Επιτροπή, η οποία ε, κατέστησε δυνατές πολυάριθμες συμβαστικές λύσεις την τελευταία εβδομάδα. Ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις εισαγωγές, ε, πεδίο εφαρμογή στόχους, αρχές. Έχουμε στον τριμερή διάλογο τελευταία φορά ε, συστήσει το θέμα των ελέγχων πολύ εντατικά, όπου πάλι βρήκαμε συμβαστική λύση όσο δύσκολο και ήταν αυτό. Ε, επίσης μπορέσαμε στον τριμερή διάλογο τελευταία φορά να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση για το πολύ περίπλοκο αυτό θέμα και χαίρομαι που από πλευράς του Κοινοβουλίου μπορέσαμε να διατηρήσουμε τις δικές μας θέσεις. Αυτό που θέλαμε ήταν κάθε χρόνο να γίνεται ε, εποπτεία, να γίνεται έλεγχος με φυσική παρουσία, με πραγματική παρουσία των ελεκτών ε, και έτσι ενώ μέχρι τώρα μόνο υπήρχε δυνατότητα, αλλά στην πραγματικότητα πολύ σπάνια μπορούσε να ε, ελεγχθεί μια ε, επιχείρηση τώρα γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, υπήρχε ζήτημα αν θα πρέπει να ανακοινώνεται αυτός ο ετήσιος έλεγχος, ο μεγάλος αυτός έλεγχος και όχι περιστασιακή, ε, προκαταβολικά ή όχι. όχι, κατά κανόνα μένουν λοιπόν απροειδοποίητη, αλλά βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και εξαιρέσεις. Ο τύπος του ελέγχου σημαίνει ότι μεταβαίνουν οι ελεγκτές και πηγαίνουν στην επιχείρηση και αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί και ανάλογα βέβαια και με την τοποθεσία της επιχείρησης να υπάρξει ε, έλεγχος. Ένα άλλο θέμα στο οποίο ε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν αυτό ε, που ορίζαν οι εντολές μας ως προς το πού θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, η Γεωργική Επιτροπή μας είχε δώσει εμάς την εντολή μας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε ε, διαφορετικές προτάσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή λύση. Στο θέμα τώρα στο οποίο δεν μπόρεσε να συμφωνήσουμε στο τριμερή διάλογο από τα πιο λεπτά ζητήματα και είναι το θέμα της επιμόλυνσης. Πώς μπορούμε να την, επι... αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να την αποφύγουμε. Είναι τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να έχει κάθε βιολογική μονάδα, κάθε βιολογική μονάδα θα πρέπει να είναι όλο και πιο σαφή, δηλαδή κανείς ε, θα πρέπει στο μέλλον να αναλαμβάνει πολύ περισσότερο την ευθύνη της λειτουργίας ε, ως προς το θέμα αυτό της εκμετάλλευσής του και βέβαια μέσα από τον τριμερή διάλογο μην συζητούμε τι είδου πιο συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να έχουμε αλλά πάντως είναι ξεκάθαρο και για μένα ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη του ελέγχου του βιολογικού τομέα παραγωγής τους, καλύτερα της προστασίας του βιολογικού τομέα παραγωγής τους, εάν ας πούμε υπάρχουν ε, ε, ζυζανιοκτώνα που χρησιμοποιούνται. Όλα αυτά είναι ευθύνη, θα πρέπει να είναι ευθύνη του κρατών μελών να εμποδίσει τη χρήση τους. Ένα ζήτημα που νομίζω ότι προκύπτει ε, τελευταία και μπορούμε να προχωρήσουμε τη Σλοβαγική Προεδρία, πιστεύω, γιατί έχουν γίνει κάποιε προκαταρκτικέ συνομιλίε. Από πλευρά του Κοινοβουλίου, εδώ και αρκετό καιρό λέγαμε ότι ουσιαστικά τμήματα του κανονισμού πρέπει να εγγραφούν στον κανονισμό βάσης και όχι σε δευτερογενή ε, νομοθετήματα ή σε ε, εκτελεστικές πράξεις. Σε αυτό δεν μπόρεσε μέχρι να καταλήξει, δεν μπορούσε μέχρι τώρα να καταλήξει το Συμβούλιο. Ε, έλεγε ότι χρειάζεται νέα εντολή για να προχωρήσει στο θέμα αυτό. Επίσης θέματα κτηνοτροφίας, θέματα σπόρων, και άλλα συναφή, ε, θα πρέπει καλύτερα να περιμένουμε να τα πιάσουμε ε, με την νέα Προεδρία του Συμβουλίου. Πάντως έχουμε προχωρήσει. Αρκετά έχουμε λύσει ζητήματα που βλέποντας τα νομίζω ότι μπορούμε να είμαι αισιόδοξο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερό. Ο, κύριος Φερό. Για το θέμα αυτό το διαπιστώσαμε και επί τόπου ότι υπάρχει μια διαφάνεια που περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις, κάτι που επιδεινώνει την, τις νέες νομοθετικές προτάσεις και πολλοί εκτροφείς έχουν πληγεί από την κρίση και στρέφονται προς τη βιολογική γεωργία, αλλά δεν έχουν αρκετές διεξόδους, ε, ούτε αρκετές επενδύσεις. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο η κοινωτική νομοθεσία σε όλες τις χώρες πολλοί γεωργοί προσπαθούν να, να διαφοροποιηθούν, να στραφούν σε πιο διαφοροποιημένες καλλιέργειες, αλλά δεν, στη, τους στηρίζει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μένουν ε, καταλελειμμένοι στη μοίρα τους, ε, οπότε καταλείπουν αυτή τη μετατροπή. Η βιολογική γεωργία είναι καλή διέξοδος, αλλά θα πρέπει να τύχουν κάποιες ενθάρρυνσεις και κάποια στήριξη αυτοί οι γεωργοί όταν αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη συμβατική υπέρ της βιολογικής γεωργίας. Κάτι που δεν συμβαίνει προς το παρόν. Ο κύριος Γιακόφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Δεν πρόκειται να εκφράσω την αισιοδοξία που εξέφρασε ο κύριος Χόισλινγκ. Εγώ διαπιστώνω ότι η φαινομενική αυτή πρόοδος επί Ολλανδικής Προεδρίας δεν με πείθει. Προοδεύουμε με πολύ αργούς ρυθμούς και αν καταφέρουμε προς τα Χριστούγεννα, δηλαδή επί Σλοβαϊκής Προεδρίας καταφέρουμε να διεκπεράσουμε αυτό το θέμα, θα ρίξω σαμπάνιες θα το γιορτάσουμε πανηγυρικά αν καταφέρουμε να το διακπεραιώσουμε έστω και στην επόμενη Προεδρία. Εγώ πολύ αμφιβάλλω πάντως ότι θα τα καταφέρουμε. Και ακόμη και αν το καταφέρουμε, διαρωτώ με αν η νέα ρύθμιση, αν ο νέος κανονισμός θα είναι πραγματικά ποιοτικός και αξιόλογος. Μήπω θα είναι απλώ κάποια καλοπιστικά στοιχεία. Δύο χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και καταλήγουμε μόνο σε κάποιες ανεπέστες αλλαγέ διακοσμητικού χαρακτήρα που δεν θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Αυτό φοβάμαι. Χαίρομαι που ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες την τελευταία φορά, έλεγχοι με βάση τον κίνδυνο. Όλα αυτά αργά κάπως κινούνται, πάντως Γενικά βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι μελιγενέστε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής παρόλα αυτά σοβαρής προσπάθειας που έγινε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά. Ο κύριος Αντρία. Ευχαριστώ. Δεν είχα α, αποφασίσει να λάβω το λόγο, αλλά με ε, παρακίνησε ο κύριος Φερά με τα σχόλιά του. Είναι τεχνικό αυτό το θέμα και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφάνεια που επισήμανε ο κύριος Φερά. Ούτε κρυπτό και παραβίστο συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Χόσλινγκ για την ενημέρωση που μας έκανε και την επισκόπηση των εξελίξεων και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την ε, Ολλανδική Προεδρία γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το θέμα, είναι τεχνικό και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια τροποποίηση του κανονισμού για τη βιολογική γεωργία. Από τη στιγμή που μιλάμε για τροποποίηση, για να θεώρηση κανονισμού, σημαίνει ότι υπάρχει υφιστάμενο κανονισμό. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την προσπάθεια και τον προηγούμενο κανονισμό. Δεν έχει κανένα νόημα η επίσπευση αν δεν ε, λαμβάναμε δεόντως υπόψη τον υφιστάμενο κανονισμό. Και συμφωνώ με τον κύριο Χόισλινγκ ότι προχωρήσαμε σε θέματα όπως ε, οι συνδυασμένες καλλιέργειες, ε, βιολογικές και συμβατικές. Επίσης ε, προχωρήσαμε σε θέματα ελέγχου. Ο έλεγχος έχει κομβική θέση στις διαπραγματεύσεις και στον κανονισμό για τη βιολογική γεωργία. Αλλά μιλούμε για 500 εκατομμύρια πολίτες που ενδιαφέρονται και εκτός από την ευρωπαϊκή αγορά έχουμε και ε, ένδο και ε, εξωτερική, διατλαντική, παγκόσμια αγορά. Γιατί έχουμε και τις εξαγωγές που θα πρέπει να προσέξουμε και εκεί υπάρχουν κάποια κατόφλια. Και για συγκεκριμένες εισαγωγές υπάρχουν ε, συγκεκριμένες διαρθρώσεις. Είναι τεράστιο το διακύβευμα αυτής της έκθεσης. Γιατί μέσω της βιολογικής γεωργίας μιλάμε για όλους τους τομείς και για όλους τους κλάδους της γεωργίας. Και είναι λογικό που προχωρούμε με αργούς ρυθμούς. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, άλλωστε είναι τόσο ευρύ θέμα και καλύπτει όχι μόνο την αδοκινοτική γεωργία, αλλά και τις ε, εταιρικέ μας σχέσεις με πάρα πολλές τρίτες χώρες. Λογικό είναι λοιπόν που καθυστερούμε. Δεν είχα προβλέψει συζήτηση για το θέμα αυτό. Προβλεπόταν μια απλή ενημέρωση από τον εισηγητή, τον κύριο Χόισλινγκ. Δεν ξέρω, κύριε Αγγιλέρη, δίστε και στο λόγο, αλλά παρακαλώ πολύ σύντομα, σε ένα λεπτό μόνο, αν γίνεται. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουμε συμφωνήσει για το θέμα των κατοφλίων. Ε, υπήρξε κάποια συμφωνία στη διαπραγματεύση για το θέμα των κατοφλίων. Μόνο αυτό θα ήθελα να μάθω. Κύριε Χόισλινγκ, εν συντομία παρακαλώ, ένα λεπτό το πολύ. Ναι. Ξέρετε την κατάσταση. Έχουμε μία πρόταση από το Κοινοβούλιο και σε αυτό είμαστε σύμφωνοι του Συμβουλίου ε, για μέτρα προληπτικά, περισσότερη ε, ανάληψη ευθύνης από τον τομέα, να, μόνο, να μην κοιτούμε μόνο μία πτυχή γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα και ε, που εξυπηρετούνται από τη βιολογική γεωργία και πρέπει να τα τονίσουμε όλα αυτά, να μιλούμε μόνο για μία ή δύο πτυχές. αλλά όπως έλεγα δεν είναι κάτι εύκολο όλο αυτό και γι' αυτό αγαπητοί φίλοι των φιλελευθέρων πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και η νέα Προεδρία φαντάζομαι ότι θα μας βοηθήσει σε αυτό. Δεν ξεκινάμε τους άλλους από μηδενική βάση. Και είπαμε ότι υπάρχει ένας ε, υφιστάμενος κανονισμός και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση μόνο. Δηλαδή έχουμε ακόμα δουλειά, αλλά δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Ευχαριστώ. Ε, συζητήθηκε Ακόμη και η κατάργηση συγκεκριμένου κανονισμού. Το θέμα είναι οι νέες διατάξεις να είναι χρήσιμες. Παρακαλώ, αν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες ή άλλες απορίες, γραπτός στείλτε mail στον κύριο Χόσλιν και εκείνος φαντάζομαι θα σας απαντήσει επίσης ηλεκτρονικά. Το πρωί είχαμε και συνεδρία των συντονιστών, αγαπητοί συνάδελφοι, και σας στείλαμε τις συστάσεις ε, των συντονιστών προς έγκριση. Δεν βλέπω παρατηρήσεις, άρα εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Οι επόμενες συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνουν στις 13 και 14 Ιουλίου. Θα έχουμε τη χαρά της δημόσιας ακρόασης με την Σλοβακική Προεδρία και τον αρμόδιο Σλοβάκο Υπουργό Γεωργίας και πολλά άλλα σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα είναι η τελευταία μας συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας πριν τις θερινές διακοπές. Ραντεβού λοιπόν στις 13 Ιουλίου. Αν προκύψει κάτι ενδιάμεσα θα δούμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο, γιατί έχουμε υψηλές προσδοκίες ε, δεδομένης της κατάστασης στην αγορά